το θέμα της ε, δυνατότητας για συλλογική δράση, επικουρικότητα βέβαια εδώ. Για να δούμε αν έχουν έρθει οι συνάδελφοι και να οργανωθούμε. Καλά, περιμένουμε μέχρι να έρθει η κυρία Γκένγκερ Ντέντεμπεργκ. και σε ακούσω την κυρία Γκαλό λοιπόν για το 30. Merci, Monsieur le Président. Alors, je rappelle euh, στους συναδέλφους οι οποίοι δεν ε, μας παρακολούσαν με μεγάλη προσοχή στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων ότι το δικαίωμα της παρακολούθησης είναι ένα αναπόσπαστο δικαίωμα των δημιουργών πλαστικών ή γραφικών έργων σε περίπτωση πνευματικών δικαιωμάτων. Κάποια κρατημέλη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι, είναι υπαρθμόν ένα στην αγορά εργοτέχνης της Ευρώπης δεν ε, παραδέχθηκαν αυτά τα δικαιώματα παρά μόνο την 1η Ιανουαρίου 12. Άλλες χώρες όπως ε, Αυστρία, Ιρλανδία και κάτω χώρες ε, εποφελήθηκαν και αυτές από τη μεταβατική περίοδο. Στις 14 Δεκεμβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση για την υλοποίηση, την εφαρμογή αλλά και τις επιπτώσεις της οδηγίας 2001 84 που αφορά αυτά τα πνευματικά δικαιώματα παρακολούθησης και αυτό αφορά και τα έργα των ζωντανών, των ζώντων καλλιτεχνών. Τα, αυτό δεν επηρεάστηκε από την ε, δημιουργία και την ε, εφαρμογή των ε, δικαιωμάτων ε, παρακολούθησης. Έγινε μια προσπάθεια να αναλυθούν οι φυστάμενες τάσεις για να διαπιστωθεί αν μπορεί να διαφανεί διαφορά ανάμεσα στις χώρες που εφαρμόζουν τα δικαιώματα παρακολούθησης και σε αυτές που δεν τα εφαρμόζουν. Πρώτη διαπίστωση, η αγορά εργών πάει πάρα πολύ καλά παρά την κρίση δεδομένου ότι το 2011 ήταν ε, χρονιά ρεκόρ με 11,57 δισεκατομμύρια δολάρια από πωλήσει έργων στην Ευρώπη. Ο όγκος των πωλήσεων επίσης αυξήθηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν εφάρμοσε τα δικαιώματα παρακολούθησης αλλά και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Δεύτερη παρατήρηση διαπίστωση μάλλον ότι η τάση έδειξε μία μετακίνηση του κέντρου βάρους της αγοράς τέχνης από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη προς τις αναδυόμενες χώρες, συγκεκριμένα την Κίνα. Στη, για την Κίνα πρόκειται για φανταστικό άλμα δεδομένου ότι είχε το 2006 το 6% της αγοράς έργων τέχνης ενώ το 2011 είχε φτάσει το 23% της, αγοράς έργων τέχνης. Βεβαίως δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τα δικαιώματα παρακολούθησης ε, για την τάση αυτή για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, οι Ηνωμένε Πολιτείε και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εφαρμόζουν τα δικαιώματα παρακολούθησης και δεύτερον γιατί η άνθηση της κινέζικης αγοράς οφείλεται στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και την εμφάνιση νέων συλλεκτών. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι η κινέζικη αγορά παραμένει περιορισμένη στους ε, εγχώριους καλλιτέχνες, δηλαδή είναι μια τοπική, τοπική αγορά που αφορά μόνο τους Κινέζους. Κατόπιν ε, μετά από αυτή την ε, αντικειμενική ανάλυση της αγοράς εργοτέχνης, το πρώτο που μπορούμε να καταλήξουμε είναι ότι από το 2001 δεν έχουμε αρνητική επίπτωση, ούτε θετική, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να, ε, να... να υπάρξουν ισόρροπες διατάξεις και αυτό να μας απασχολήσει ώστε η, η κατάσταση να είναι ισόρροπη Χάρη στη μείωση των ποσοστών που ισχύουν. Το ανώτατο όριο, σας θυμίζω, είναι τα 12.500 ευρώ, όχι πάρα πολύ ψηλό. Υπενθυμίζω επίσης ότι οι μικρές πωλήσει εξαιρούνται, αποκλείονται και μια πολύ σημαντική διάταξη είναι η φορολογική απαλλαγή της πρώτης μεταπόλησης για τον πρώτο αγοραστή. Πρέπει να σκεφτούμε και να γνωρίζουμε ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Κίνα και αυτές ε, ενδεχομένω σκέφτονται την εισαγωγή του δικαιώματος παρακολούθησης γιατί ε, τα έργα τέχνης αυτού του είδους ε, συνεπάγονται μεγάλες περιόδους αναμονής για τους καλλιτέχνες μέχρι ότου κερδίσουν ε, χρήματα. Και αυτό είναι ένα θέμα που και εμάς μας απασχολεί. Οι χώρες που ανέφερα και τελευταίο το Ηνωμένο Βασίλειο ε, έθεσαν σε εφαρμογή αυτή την οδηγία την 1η Ιανουαρίου 2012 σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε κάποια απόσταση ώστε να μελετήσουμε τον αντίκτυπο αυτής της οδηγίας του 2001. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη 2014 ως χρονιά επαναξιολόγησης και εγώ στην γνωμοδότησή μου ζητώ να μελετηθεί συγκεκριμένα το ποσοστό που ισχύει και οι κατηγορίες των δικαιούχων γιατί υπάρχουν και οι ιδιοκτήτες γκαλερί κλπ. Αυτά όσον αφορά αυτή την έκθεση. Τώρα, όσον αφορά την κατάθεση τροπολογιών, προτείνω την 7η Σεπτεμβρίου ως ε, προθεσμία. Και φυσικά είμαι στη διάθεση των συναδέλφων να ακούσω τις απόψεις τους. Ευχαριστώ. Τέιλορ, παρακαλώ. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Γκάλο για μια πολύ συνοπτική έκθεση και συμφωνώ με αυτά που είπε στο, στην έκθεση του ότι τα στοιχεία είναι ότι ε, δεν έχουμε αρνητικές επιπτώσεις από το δικαίωμα παρακολούθησης. Επειδή όμως η οδηγία εφαρμόστηκε μόνο τον Ιανουάριο του 2012, συμφωνώ με την πρόταση να επανεξεταστεί ο αντίκτυπος το 2014. Επειδή παγκοσμιοποιείται η αγορά έργων τέχνης όπως μας εξήγησε η κυρία Γκάλο, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τη μελέτη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, να γίνουν διαπραγματεύσεις ώστε να υπάρχει ένα άρθρο 14β της Σύμβασης της Μόνης, το οποίο να είναι υποχρεωτικό. Ένα δευτερεύον θέμα σε σχέση με το σημείο 15 της έκθεσης της κυρίας Γκάλο είναι ότι θα πρέπει ίσως η Κομισιόν να επανεξετάσει το ανώτατο όριο όπως επίσης και τα, ε, τα, τα ποσά που ε, ισχύουν. Άλλα σχόλια παρακαλώ. Η κυρία Γκάλο από ό,τι βλέπω ε, νεύει καταφατικά, είναι ικανοποιημένη, δεν υπάρχει ποτέ άλλο να προσθέσει. Θέλετε κάτι άλλο κυρία Γκάλο. Διαπιστώνω ότι είναι ένα θέμα που δεν ε, κάνει, ε, συγκεντρώνει το μεγάλο ενδιαφέρον, δεν προκαλεί το πάθος στους συναδέλφους. Αυτά. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Ε, θα πρέπει να δούμε και, τους, και τις τροπολογίες 7 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Κλείνει το θέμα αυτό και πάμε στο 29. Έχουμε τον κύριο Τσιεύκα, έχουμε την κυρία Γκερίνγκερ. Δε Ödenberg. Έχετε το λόγο, κυρία Γκερίνγκερ Δε Ödenberg. Παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έχει να κάνει βέβαια με επικουρικότητα. Λοιπόν, ε, ε, φέτος το Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της ε, για κανονισμό του Συμβουλίου που έχει να κάνει με την εξασφάλιση του δικαιώματος για συλλογική δράση σε περίπτωση παραβίαση του δικαιώματος για κατάσταση και παροχή υπηρεσιών. Πρόκειται για την πρόταση τη δύο δηλαδή. Η νομική βάση ήταν το άρθρο 353 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαίνεται να συμφωνεί και το Συμβούλιο ε, φαίνεται να αναμένεται ότι θα συμφωνήσει και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ε, το πρωτόκολλο 2 της Συνθήκης Λισαβόνας προτείνει τη δυνατότητα για τα ε, κοινοβούλια των κρατών μελών να θεωρήσουν τα μέτρα αυτά και να ε, παρουσιάσουν μια αιτιολογημένη γνωμοδότηση εφόσον θεωρούν ότι το προτινόμενο κείμενο δεν συμφωνεί, δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Εάν πάνω από τα μισά κοινοβούλια των 100 μελών διατυπώσουν τέτοια πρόταση, τότε θα πρέπει να αναθεωρηθεί η εν λόγω ε, πρόταση κανονισμού, είτε να τροποποιηθεί το κείμενο, είτε να ε, αποσυρθεί τελείως. Είναι η λεγόμενη διαδικασία της κίτρινης κάρτας. Έχει ήδη τέτοιο προηγούμενο ε, λάβει η χώρα. Στην δε διαδικασία υπάρχει μια απλή λύση. Εάν η απλή πλειοψηφία των Εθνικών Κοινοβουλίων δώσει αρνητική γνωμοδότηση, θα πρέπει το θα πρέπει η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου να εξετάσει αν είναι σύμφωνη με την αρχή της επικορικότητα ή προτινόμενη από την Επιτροπή Νομοθετική Πράξη. Εάν ε, δεν συνάδει με την αρχή της ε, επικουρικότητας, τότε ισχύει τότε θα πρέπει να αποσυρθεί. Και υπάρχει και η, η διαδικασία της κόκκινης κάρτας τότε, οπότε συμβαίνει το εξής. Οχτώ εβδομάδες μετά τη γνωμοδότηση που έληξαν στη δική μας την περίπτωση στις 26 Μαΐου και έτσι προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Συμβούλιο των Επιτρόπων, το συλλογικό όργανο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να συζητήσει στην προσοχή του συνεδρίαση το ε, κείμενο αυτό, τη γνωμοδότηση δηλαδή να την υποστηρίξει, οπότε μπορούν να ληφθούν σχετικές αποφάσει. Να δούμε πώς διαμορφώνεται δηλαδή η σχετική η, η κατάσταση. Το άρθρο 38α του κανονισμού προβλέπει ότι η μη αιτιολογημένη γνωμοδότηση οι γνωμοδοτήσεις, ε, μη αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων πρέπει να καλύπτουν, να είναι τουλάχιστον το 1 τρίτο των ανετικών γνωμοδοτήσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Τη συνέχεια την ορίζει το άρθρο 76 συνθήκη ε, για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ω εκ τούτου θεωρώ ότι ε, δεν έχουμε περιθώρια επιλογή και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τι συστάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλοί είναι οι περιορισμοί που εισάγει το έγγραφο αυτό, πολλέ είναι οι αντιδικίε με τα κράτη-μέλη, τα σημεία στα οποία διαφωνούμε και επομένως θα πρέπει να μεριμνήσουμε η νομοθετική πρόταση να συμφωνεί με την αρχή της επικουρικότητας. Περιμένουμε από την Επιτροπή και πιστεύω ότι κατά την προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα έχουμε στη θέσή μας το έγγραφο αυτό, αλλά όπως και να έχει Δε και ένα μήνα δεν έχουμε πάρει πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή περιμένουμε καλύτερα μέχρι το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το προτιμότερο. Ευχαριστώ πολύ, Ταντέους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ του Άξελ Βος ε, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ε, δική του την άποψη για το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε η Λίντια Γκέριγκερ. Πρόκειται για ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον και από πλευράς νομικής βάσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπε και η Λίντια, πρότεινε ως νομική βάση το άρθρο 352. το άρθρο δηλαδή που περιλαμβάνει τη ρήτρα της ευελιξίας, της ελαστικότητας και είναι δύο τα στοιχεία που ενδιαφέρουν το συγκεκριμένο άρθρο και θα ήθελα να τα επισημάνω για να εξηγήσουμε ακριβώς και πώς εφαρμόζεται αυτή η νομική βάση. Πρώτον, εάν οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρηθούν απαραίτητες ώστε να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τους στόχους και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνθήκη δεν προβλέπει να, μην, ε, να ληφθεί συγγνώμη, κάποια συγκεκριμένη δράση, το Συμβούλιο ομόφωνα επί τη βάση προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να το κάνει. Αυτά εγκρίνονται συνήθως με μια ιδιαίτερη διαδικασία πάντα βάσει πρόταση τη ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, με επικύρωση του Κοινοβουλίου. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, στα πλαίσια της διαδικασία ελέγχου και της αρχής της επικουρικότητας, στο άρθρο 5 παράγραφος 8 της Συνθήκης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί την απόφαση ενεργοποίησης αυτής της ρήτρα ε, στα Εθνικά Κοινοβούλια. Εάν λοιπόν πρέπει να βασιστούμε στο κείμενο όπως είναι γραμμένο και το ε, κλάβουμε κατά γράμμα δεν υπάρχει κανένα θέμα συζήτησης. Αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ δύο πτυχές. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρκετά αμφίσιμη ε, στο κείμενό της. και δεν φαίνεται να αιτιολογείται η εφαρμογή του εν λόγω άρθρου για έναν πολύ απλό λόγο. Το άρθρο αυτό έχει προβλεφθεί για τις έκτακτες περιπτώσεις, τις εξαιρετικές περιπτώσεις, τις οποίες δεν υπάρχει ε, άλλη διέξοδος, δεν υπάρχει δεύτερη εναλλακτική λύση. Μέχρι του δε το άρθρο αυτό ε, στο πρόσφατο χρονικό διάστημα ε, χρησιμοποιήθηκε μόνο μια φορά. Είχαμε μια έκθεση, την έκθεση Ζόμπρου, που αφορούσε την επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφορά μεταξύ της συγκεκριμένη περίπτωσης και της ε, περίπτωσης που συζητούμε τώρα είναι γνωστή και νομίζω ότι είναι και προφανής. Σε εκείνη την περίπτωση πρόκειται για ένα καθαρά τεχνικό ζήτημα, ενώ εδώ συζητάμε ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά πολιτικό. Η ρήτρα λοιπόν αυτή τη ευελιξίας ε, ε, του άρθρου 352 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ε, η έσχατη λύση στην περίπτωση στην οποία δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι ε, όροι από πλευράς συνθήκης ε, και δεν καθορίζεται κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία για να επιτευχθεί κάποιος στόχος. Η πρόταση λοιπόν του κυρίου Βος είναι η εξής. Βάσει του άρθρου 37.3 του ιστορικού κανονισμού μας, η, Ευρωπαϊκή, η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων μπορεί να λάβει νομικά μέτρα. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια αποφασίσει να ξεκαθαρίσει τη θέση της, κάτι το οποίο δεν έχει κάνει μέχρι τούδε. Αν αποφασίσει λοιπόν να τροποποιήσει ή να αναστείλει την απόφασή της, πάντα παραπόμποντας ε, στο άρθρο 352, ο κύριος Φως προτείνει η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να ετοιμάσει έκθεση πρωτοβουλίας η οποία θα εξετάζει κατά πόσο είναι κατάλληλη η νομική βάση ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι κατάλαβα από τις δύο παρεμβάσεις θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή εδώ εκπροσωπείται. Είναι κάποιος ε, που μπορεί να αναλάβει να μας μιλήσει εκ μέρου επιτροπή. Ή τη Επιτροπής ή δεν προτιμάει να τοποθετηθεί η Επιτροπή προς το παρόν. Όχι από ό,τι φαίνεται. Κάποτε θα πρέπει. Α, θέλετε να μιλήσετε, μάλιστα. Ναι, ευχαριστώ, πολύ. πολύ. Νομίζω ότι ήδη έχει υποθεί ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι εδώ με μια άνευ προηγουμένου υπόθεση από τη θέση εφαρμογή της συνθήκης της ε, Λισαβόνας με πολύ μεγάλο πολιτικό αντίκτυπο. Είναι σαφέστατο ότι οι διατάξεις αυτές έχουν σταγματική βαρύτητα, σταγματική αξία και ε, σχετίζονται με τις νέες εξουσίες που δίνονται και αναγνωρίζονται στα εθνικά κοινοβούλια ως προς την αρχή επαλήθευσης της ε, επικουρικότητας. Άλλωστε αυτό έχει δηλωθεί και από την ε, ομιλία του κυρίου Μπαρόσο στην ε, τελετή θέση ισχύ της συνθήκης Λοιπόν, το, η Επιτροπή Συλλογικό Όργανο επιβεβαίωσε το Μάιο ότι η διαδικασία της κίτρινης κάρτας έχει τεθεί σε λειτουργία. Γιατί 19 ψήφοι από τις, τις 54 ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων, ε, εν, μία ψήφος παραπάνω από τις 18 που είναι το όριο για την εκείνη τη και άρα προτείνεται η δυνατότητα είτε της διατήρησης είτε της απόσυρσης είτε της τροποποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ε, νομοθετικής πρότασης. Αυτή τη στιγμή έχουμε διεξοδική ε, μελέτη των συνθήκων, των όρων. Είναι θέμα βεβαίως στα εθνικά κοινοβούλια, πολύ σημαντικό, με πολύ μεγάλη πολιτική βαρύτητα και καθώς καταλαβαίνετε δεδομένης χρονικής στιγμής ε, δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες ενδείξεις. Θα πρέπει να προχωρήσουμε. Μάλιστα, άρα έχετε πολλή δουλειά για το καλοκαίρι, έτσι, παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, θεωρώ και το έχω ξαναπεί ότι η αρχή τη επικουρικότητα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα από τη δική μα Επιτροπή. Πολλοί από εμά, του φιλελεύθερου, αλλά και από άλλε πολιτικέ ομάδε, στον ε, στον προεκλογικό μα αγώνα υπογραμμίσαμε ιδιαίτερα τη μεγάλη σημασία και το σεβασμό που σκοπεύουμε να δείξουμε στην αρχή τη επικούρικότητα. και λέγαμε ότι θα πρέπει να ρυθμίζονται μόνο τα θέματα ε, που ρυθμίζονται κατά καλύτερο τρόπο από το ευρωπαϊκό επίπεδο και όλα τα υπόλοιπα στο εθνικό, το τοπικό, το περιφερειακό όπω πρέπει. Τρία χρόνια πέρασαν και ήρθε τελικά το θέμα τη επικούρικότητα με πολύ μεγάλη ενάργεια μπροστά μα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία και να πούμε ότι ιδιαίτερο πρόβλημα μπορεί να είναι το ότι δεν έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία στα κράτη-μέλη, δεν έχουν δηλαδή μέχρι στιγμή ε, ε, αναπτύξει επαρκή ε, εργασία, επαρκέ έργο τα κράτη-μέλη, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε περιφερειακό και οι περιφέρειε ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει αυτή τη δουλειά που θα έπρεπε τη συνεργασία μεταξύ του. Ε, Επίση πρέπει να διαπιστώσουμε ότι όταν και εάν πράγματι θέλουμε να έχουμε ένα πολιτικό αποτέλεσμα σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν θεωρείτε ότι είναι σημαντικό κάτι δεδομένη της κρίση για το του ευρώ, δεδομένη τη χρηματοοικονομική κρίση, βλέπουμε ότι πάντοτε βρίσκεται η κατάλληλη νομική βάση και δίνονται οι λύσει χωρί προβλήματα. Άρα βρίσκεται πάντα ο πολιτικό τρόπο να βγούμε από το αδιέξοδο. Και άρα θα πρέπει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα να κοιτάξουμε το θέμα αυτό, την επίκριση δηλαδή τη αρχή τη επικουρικότητα. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με του συζητητέ ότι ε, εφόσον προβλέπεται από τη συνθήκη, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και δεν νομίζω θα σα ξαφνιάσει ύστερα από τρία χρόνια της λειτουργίας συνθήκη, δεν χρειάζεται να περάσει μήνε για να επαληθεύσει το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει μέχρι το Σεπτέμβριο να μα έχει έτοιμη στην προσεχή μα συνεδρία τη Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων μία έκθεση για τι θέσει τη Και θα ήθελα να συμφωνήσω με το όσοι είπε ο Εάν δεν ε, το πράξει η Επιτροπή, θα πρέπει να λάβουμε εμεί να προξενήσουμε αυτή τη διαδικασία. Καλώ λέει ο πρόεδρο. Νομοδότη το Σεπτέμβριο θα έχετε δύο μήνε περιθώριο από την Επιτροπή, επομένω δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα τα καταφέρετε. Καλώ αφήνουμε το θέμα αυτό. Δεν κανεί άλλο το λόγο. Και πάμε στο σημείο 30. Την άλλη έκθεση τη κυρία Γκαλό, προσωπικά δεδομένα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι η συγγήτρια για γνωμοδότηση μιας, ε, για σύνταξη μάλλον μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας, για γνωμοδότηση πάνω σε μια νομοθετική πρωτοβουλία που είναι σημαντική σε δύο επίπεδα. Καταρχάς και το γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς ειδικά, τη, δεδομένη της ε, ε παρουσίας ε, των μέσων του ίντερνετ των πληροφοριών που διακινούνται μέσω του ίντερνετ ε, παντού, που μπορεί κανείς να βρει μέσα από ένα μηχανισμό ε, αναζήτησης ε, του διαδικτύου, που δίνουν στον πολίτη την αίσθηση ότι δεν είναι προστατευμένα τα προσωπικό του δεδομένα και που άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς για να έχουμε ψηφιακό περιεχόμενο σοβαρό και ανταγωνιστικό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενθυμούμενοι βέβαια και τον μεγάλο αδελφό του ε, Orwell ότι ο μεγάλος αδελφός πλέον δεν είναι τα κράτη, δεν είναι τα μεγάλα κράτη αλλά ο, ο πάροχος ε, ψηφιακού περιεχομένου που βλέπουμε πάντα κρυμμένο πίσω από υποθετική διαφήμιση, από διάφορα μηνύματα κτλ. Αυτή η προστασία λοιπόν των προσωπικών δεδομένων εγγράφεται μέσα σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης, μια συζήτηση που έχει να κάνει με την ανάπτυξη και της ψηφιακής οικονομίας. Η προστασία λοιπόν των προσωπικών δεδομένων βεβαίως πρέπει να είναι αποτελεσματική, αλλά πρέπει να είναι και αναλογική ώστε να μην παρεμποδίσει την ανάπτυξη αυτών νέων υπηρεσιών και προϊόντων που θα αποβούν ε, εις όφελος και συμφερόν των ε, πολιτών. Ταυτόχρονα αυτή η νέα ψηφιακή οικονομία θα πρέπει να είναι συμβατή και με τις λοιπές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί παραδείγματι τη στρατηγική για την ε, για το cloud computing, για την λειτουργία του νεφελώματος στο διαδίκτυο και για άλλα αντίστοιχα ζητήματα. Ε, συζητήσαμε την έκθεση πρωτοβουλίας ε, του Άξελ Φως με μια ιδέα για μια συνολική ε, προσέγγιση. Λαμβάνω υπόψη την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας και την πρόταση που, της Επιτροπής που έχει υιοθετήσει το Κοινοβούλιο. Η αρχή της Οδηγίας 95 που αποτελεί το κείμενο αναφορά εν προκειμένου παραμένει επίκαιρη. Και αυτή είναι και η πρόταση για την οποία η πρόταση του κανονισμού ενισχύει, διατηρεί αυτές τις βασικές αρχές αλλά και διαφυλάσσει και ενισχύει τα δικαιώματα των χρηστών. Ένα μήνυμα λοιπόν σαφές από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο μας ικανοποιεί και όπου θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν ε, πρέπει να λησμονήσουμε ότι πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ναι, μένα, σε αυτά αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο, αλλά ταυτόχρονα και δεδομένα εκτός ε, εκτός σύνδεσης, δηλαδή offline, που παραμένουν πάρα πολύ σημαντικά. Χαρακτηριστικό που παραμένει πολύ σημαντικό. Επομένως, θα πρέπει να συζητήσουμε τι σημαίνει δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει και σήμερα αλλά και για το μέλλον. Βλέπω μία μόλις ώρα είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με ειδικού του, ψηφιακού περιεχομένου που μου εξήγησαν παραδείγματι ότι είναι κορεσμένες πλέον οι διευθύνσεις IP και ότι δεν θα υπάρχουν νέες, δεν θα μπορούμε δηλαδή να χορηγήσουμε νέες διευθύνσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν μέχρι και 100 χρήστες πάνω στην ίδια ε, διεύθυνση IP. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πρόκειται αυτή τη στιγμή για ένα προσωπικό, προσωπικού χαρακτήρα δεδομένο, αλλά μπορεί αύριο, όταν θα είναι κορεσμένο αυτό ο χώρο, να μην ε, είναι πλέον προσωπικό δεδομένο. Ε, άρα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα του ορισμού μα. Δεύτερον, και αυτό προτείνουν και τα κείμενα, την προστασία των ε, δεδομένων από τον προσδιορισμό τη επεξεργασία οι οποίε μπορούν να τύχουν, δηλαδή το άρθρο 23. Συμφωνώ απόλυτο σε αυτό. Από την άλλη όμω, σε σχέση με την παράδοση υπαριθμών 2 του άρθρου 23, μου γινόνται πολλά, πολλά ερωτηματικά γιατί προτείνει μια ε, αυτοδύναμη προστασία, ενώ υπάρχει στην παράγραφο 13 ο κανόνας για ελαχιστοποίηση των δεδομένων, που λέει δηλαδή ότι τα δεδομένα θα πρέπει να μειωθούν στο απολύτως απαραίτητο ελάχιστο, που αντιστοιχεί στο στόχο της χρήσης τους. Επομένως, η προστασία ε, η αυτεπάγγελτη προστασία δεν καταλαβαίνω τι λόγο έχει όταν περιορίζεται στο ελάχιστο η ε, παροχή των στοιχείων. Αλλά ίσως κάποιος να μου το εξήγησε. Και άλλο τελευταίο σημείο που είναι ίσως και το πιο γνωστό από την κοινή γνώμη, είναι το, το στοιχείο το σχετικό με το δικαίωμα στην ψηφιακή λύθη που προτείνει το άρθρο 17, όπου και πάλι θα πρέπει να αποφύγουμε τις ε, τις προτάσεις τις ε, πιο εθερβάμονες, γιατί πάλι μιλώντας με ειδικού του ψηφιακού περιεχομένου, αντιλαμβάνομαι ότι απόλυτη διαγραφή του, ε, του ψηφιακού υλικού είναι μάλλον αδύνατο να επιτευχθεί και ως εκ τούτου το δικαίωμα στη λύθη είναι δικαίωμα μεν, αλλά δεν ισοδυναμεί με δικαίωμα στην απόλυτη απάλληψη των στοιχείων. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Με συγχωρείτε, αλλά σήμερα παραμίλησα. Και το τέταρτο σημείο αφορά την συνένεση. Είναι πολύ σημαντικό η συνένεση να αποτελεί ε, συστατικό στοιχείο της νομιμότητας τη επεξεργασία των στοιχείων αυτή τη συνένεση. Η συνένεση δεν μπορεί να είναι σιωπηρή που δεν είναι, αυτό είναι σαφέ. Άρα θέλουμε ρητή συνένεση. Συνένεση η οποία απορρέει από σαφή και λελογισμένη βούληση μπορεί όμως να εκφράζεται μόνο με την ε, υπόδειξη ενός σημείου σε ένα τετραγωνάκι και πάλι συμφωνώ με την αρχή της ρητής συνένεσης πλην όμως ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η αρχή με τρόπο ευφυή ώστε να μην επιβαρύνονται με υπερβολικές, ε, υπερβολικά αυστηρές διατάξεις και υποχρεώσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ενδεχομένως δεν θα είχαν τη δυνατότητα να, συγγνώμη, να ε, ανθέξουν το βάρος τέτοιων υπερβολικών υποχρεώσεων. Και επίσης ο υπεύθυνο επεξεργασίας έχει υποχρέωση μέσου και όχι αποτελέσματος. Πρέπει να θέσει σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα ε, μέσα, όλες τις απαραίτητες τεχνικές δηλαδή δυνατότητες που υπάρχουν. Επίσης, τελευταίο και σημαντικό σημείο, προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, των ανελίκων, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό πιστεύω όλοι συμφωνούμε. Ένα έκτο σημείο πολύ σημαντικό και που χρειάζεται διεξοδική ανάπτυξη αλλά θα σας απαλλάξω σήμερα γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να το ξαναδούμε άλλη φορά το θέμα διεξοδικότερα, έχει να κάνει με την διαβίβαση δεδομένων προς, τρίτα χρόνια, προς τρίτες χώρες, γιατί γνωρίζουμε βέβαια ότι το ίντερνετ έχει καταργήσει τα σύνορα και ως εκ τούτου ο έλεγχος θα πρέπει να ασκείται ε, δυνάμει των άρθρων 40 και επομένων όπου προβλέπεται ευελιξία ως προς τους μηχανισμούς που οδηγούν σε ένα επίπεδο, όπως ονομάζεται, κατάλληλης ή δέουσας προστασίας. Ορίζονται κριτήρια και προϋποθέσεις ε, για την έγκριση από την, Επιτροπή μιας διαπίστωσης ε, δέουσας προστασίας. Το άρθρο 42 δε υπάγει αυτήν την ε, έγκριση σε περίπτωση απουσίας απόφασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ύπαρξη κατάλληλων εγγύσεων όπως ονομάζονται, δηλαδή με κάποιες ρήτρε τύπου, ε, τυπικές, για τις επιχειρήσεις, ε, δηλαδή δεσμευτικές ε, ρήτρε που μπορούν σε μια άλλη περίπτωση να είναι και να υπάγονται σε κάποιες συγκεκριμένες και δεσμευτικές προϋποθέσεις. Χρονοδιάγραμμα. Στο χρονοδιάγραμμα μπορούμε να εξετάσουμε, πιστεύω, την ε, πρόταση για γνωμοδότηση στην προσεχή μας συνεδρία του Σεπτέμβριο, οπότε και μπορώ να σας δώσω τις περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τροπολογιών και τη σχετική προθεσμία. Πρόεδρε, ευχαριστώ και με συγχωρείτε γιατί θα πρέπει να σοπάσω. Τώρα έχει κλείσει η φωνή μου πια. Κυρία Γκαλό, ευχαριστώ. Πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα. Έχετε το λόγο. Η κυρία Τσέιλορ. Πολύ σύντομα, θα ήθελα απλώς να πω ότι στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε, με όλα τα δεδομένα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όπως ανέφερε και η κυρία Γκάλο, ε, το θέμα αυτό και η προστασία των δεδομένων αφορά όλους. Γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα προστατεύσουμε την ιδιωτική ζωή του καθενός και να επιτρέπουμε ταυτόχρονα να υπάρχουν ε, οι υπηρεσίες που βασίζονται στο διαδίκτυο και καινοτομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εξετάσουμε διότι ε, αναπτύσσεται συνεχώς η τεχνολογία και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε νομοθεσία που να μπορεί να προσαρμόζεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Αυτό αφορά και τους χρήστες αλλά και όσους παρέχουν υπηρεσίες δεδομένων και προσβλέπω στη συνεργασία με την κυρία Γκάλου για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κυρία Λίχτενμπέργκερ. Πρόεδρε ευχαριστώ για την πρώτη αυτή έκθεση την κυρία Γκαλό. Όντως είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα αλλά δυστυχώς δεν ήταν τόσο διεξοδική και σαφής η λύση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή της, όπως θα έπρεπε κανείς να περιμένει, ε, έτσι ώστε να μπορούν οι αρχές οι αρμόδιες για την προσοχή των προσωπικών δεδομένων να κάνουν ουσιαστική δουλειά. Εν πάση περιπτώσει όμως έχουμε εδώ να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια ζητήματα και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το εξής ότι θα πρέπει να είμαστε θέση να ε, προβλέψουμε ενδεχόμενε μελλοντικέ εξελίξει, ε, πράγμα το οποίο είναι αδύνατο. Μίλησε η συνάδελφο Φερρυπίν για το νεφέλωμα, το cloud, ε, κάτι το οποίο μπορεί να έχει τεράστιες δυνατότητες να προσφέρει, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλες προκλήσεις λόγω παραδείγματι της χρήσης επαγγελματικού χαρακτήρα δεδομένων. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό οι cloud computing strategies θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ μεγάλη προσοχή αν είναι κατάλληλε για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, ναι ή όχι. Επίση, ένα θέμα θα πρέπει να είναι αν χρειάζεται ευρωπαϊκή υποδομή από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή ε, εξαρτώμαστε μόνο από αμερικανικό server. Θα πρέπει να ε, ομολογήσουμε, όσο δεν υπάρχουν δηλαδή ευρωπαϊκοί servers, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν υπάρχει θέμα προστασία προσωπικών δεδομένων, γιατί είναι πάνε όλα τα δεδομένα στου ε, ΗΠΑ και ο Ευρωπαίο πολίτη εξαρτάται από την βούληση των αρχών εκεί. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Άλλες παρατηρήσεις για τα ερωτήματα που ετέθησαν που βεβαίως και με τροπολογίες θα διευκρινίσουμε. Η προϋπόθεση για διαφάνεια, η απέτηση για διαφάνεια είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα ασφαλώς. Αλλά δεν μπορεί να μας εμποδίσει αυτή η υποχρέωση διαφάνειας να βρούμε λύσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν ε, μια διαφορετική, ένα διαφορετικό δρόμο, μια παρέκκληση ούτως υπήν μικρομεσαίε επιχειρήσει. Μικρομεσαίε επιχειρήσει χαρακτηρίζονται αυτέ που έχουν ε, κάτω από 250 ε, εργαζομένου Εκεί πέρα ήδη υπάρχουν προβλήματα και, γιατί δεν νομίζω, πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο κριτήριο αριθμό των εργαζομένων μια επιχείρηση. Ε, πρώτον, διότι σε αυτό το τομέα τη επιχείρηση θα πρέπει να δούμε ότι μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλέ επιχείρησει οι οποίε αποθηκεύουν, ε, αποθηκεύουν υπηρεσίες αποθηκεύει μάλλον υλικό συγγνώμη, σε ε, παρόχους υπηρεσιών και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τις αρχές αυτές, τις συγκεκριμένες αυτές επιχειρήσεις και άρα δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα η οποιαδήποτε ρύθμιση προτεθεί. Ε, μπορεί να υπάρξει διάσπαση επί παραδείγματι σε διαφορετικές αρχές προστασίας των δεδομένων. Ε, για την Αυστρία μόνο μπορώ να σας πω ότι ε, μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα πέντε διαφορετικές αρχές προστασίας των δεδομένων συναρμόδια σε περίπτωση τέτοιας εξωτερική αποθήκευση δεδομένων και εδώ το κριτήριο δεν μπορεί να είναι μόνο ο αριθμό των απασχολουμένων αλλά άλλα συγκεκριμένα στοιχεία και εδώ πέρα ακριβώς θα θέλω να επισημάνω ότι είναι εσφαλμένη η προσέγγιση του ζητήματος από τη σκοπιά του αριθμού των εργαζομένων. Μπορεί να υπάρχουν ε, και άλλα κριτήρια όπως ο κύκλος εργασιών λοιπά Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις με 30-50 μόνο εργαζομένους αλλά με τεράστιο κύκλο εργασιών. Ε, για την ε, περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική και θα ήθελα να είμαστε θα ήθελα να προταθεί μια λύση ενός πάρα πολύ αυστηρού opt-in ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος να παραβλέψει μία ε, παρατήρηση σε μια σελίδα συμβολέου, αλλά να πρέπει ε, ε, ρητά και ηθελημένα να δεχθεί να βιβάζονται τα στοιχεία του. Αυτό είναι το opt αυτή είναι η μόνη δυνατότητα που βλέπω να αριθμιστεί το θέμα ουσιαστικά. Δεν έχω εγώ προσωπικός ποτέ δεχθεί, δεν ξέρω ποτέ να έχω δεχθεί να ε, διατεθούν τα στοιχεία μου σε κάποιον άλλο για εμπορικό σκοπό κτλ. Παρόλα αυτά όμως ε, λαμβάνω στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο χιλιάδες μηνύματα είτε για ε, σπα είτε για κέντρα αδυνατίσματος είτε για ό,τι άλλο και πάση περιπτώσει διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει προστασία των προσωπικών δεδομένων και ασφαλώς κάποιος μπορεί να ανοίξει τον τηλεφωνικό κατάλογο και να πάρει τα στοιχεία αυτά τηλέφωνο και το καθεξής και να ενοχλεί τους ε, πολίτες. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί να διατεθούν τα προσωπικά δεδομένα χωρίς ποτέ να έχει δώσει συνένεση ο ε, ενδιαφερόμενο πολίτη και τι πολλέ φορέ αυτέ οι επιχειρήσεις έχουν δεσμευτεί ρητά να μην διαβιβάσουν ε, τα στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με το opt-in λοιπόν θα πρέπει να ε, αντιμετωπιστεί για το ζήτημα του δικαιώματο στη λύθη, ε, right to be forgotten. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ απόψει. Κάποιοι θέλουν μια πάρα πολύ ε, διασταλτική ερμηνεία της υπόθεσης αυτής. Ε, που θα μπορούσε να οδηγήσει όμως σε προβλήματα ως προς την ε, εφαρμογή των διατάξεων ή την ε, ανάπτυξη, την λειτουργία διαδικασιών, ενδεχομένως δε και νομικών αγώνων, σε περίπτωση όπου δεν διατίθενται πλέον τα στοιχεία αυτά. Αλλά από την άλλη υπάρχει και η αρχή της υποχρέωσης για πρόνοια, για προστασία, diligence εν προκειμένου. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικό λοιπόν και να πούμε ότι πρέπει να δοθεί μια δυνατότητα να σβήσει κανείς με τρόπο υπεύθυνο και διεξοδικό τα δεδομένα του χωρίς περιορισμούς που πιστεύω μπορεί να εξασφαλιστεί με μια ρύθμιση που θα λέει που θα ορίζει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα επιτυγχάνεται αυτή η απάλληψη των στοιχείων. Κάθε πολίτης, κάθε ιδιώτης έχει το δικαίωμα να επιλέξει να διαγράψει τα στοιχεία του από το διαδίκτυο. Επίσης, κάτι άλλο που σημείωσα, καθοριστικό και αποφασιστικό σημείο θα είναι ε, η πρόταση για τη συνολική προστασία των δεδομένων, διότι θα πρέπει να είναι δυνατό να γίνεται η επαλήθευση προκαταβολικά όλων των στοιχείων. Δηλαδή, εάν δεν ε, συμπεριλάβουμε επιπλέον λειτουργίες, μπορεί κανείς προκαταβολικά να είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσει την, ε, το φόρτο εργασίας που μπορεί να φέρει η λειτουργία ενός ε, κανονισμού μιας διατάξεως. Εάν όμως εισαχθούν πολλές άλλες προϋποθέσεις, τότε η κατάσταση περιπλέκεται σημαντικά. Αυτό ήθελα να επισημάνω. Δεν βλέπω τίποτε άλλο ουσιαστικά να προσθέσω. Χρήσιμο τουλάχιστον. Σημαντικό πρόβλημα βεβαίως θα είναι το ζήτημα της διαβίβασης τρίτα κράτη προσωπικών δεδομένων και υπεξεργασία δεδομένων από τρίτα κράτη. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά εν πάση να μπορέσουμε καν να το λύσουμε, αλλά εν πάση εκεί που έχει αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, επιβάλλει την ε, λειτουργία αυτών των διατάξεων, διότι αν αφήσουμε ένα τεράστιο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας για τα κράτη-μέλη, η να αφήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τεράστιο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας για τα κράτη-μέλη, τότε ουσιαστικά εξουδατερώνεται το νόημα όλης αυτής της προσπάθειας και παρακαλώ να προσέξουμε ιδιαίτερως να κάνουμε ένα ε, νομοθέτημα το οποίο θα είναι εφαρμόσιμο εύκολα, θα έχει ένα λογικό περιθώριο ε, ευελιξίας για θέματα διεθνή ή διεθνικά, χωρίς όμως υπερβολική χαλαρότητα, γιατί τότε θα ακυρωθεί όλο το νόημα της προσπάθειας. Ε, ένα παράδειγμα που μπορώ να σας δώσω είναι το πολύ επίκαιρο στη Γερμανία ζήτημα της νομοθεσίας για την ε, ανακοίνωση προσωπικών δεδομένων πολιτών που μπορεί από το ένα κρατήδιο της Γερμανίας στο άλλο να διαβαστούν από εμπορευομένους κτλ. Ε, φανταστείτε τώρα να ε, ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το ένα κράτος στο άλλο να επιβάλλονται εξαιρέσει επί των εξαιρέσεων και να καταστεί ε, τελείως ανεφάρμοστη όλη αυτή η νομοθεσία. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ κυρία κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, πιστεύω, ότι τα προσωπικά μας δεδομένα πλέον αποτελούν αντικείμενο αγοράς. Ότι όχι μόνο συγκεντρώνονται, φυλάσσονται, συλλέγονται, αναλύονται, ε, αρχιοθετούνται, αλλά πολλούνται και αγοράζονται. Πράγμα που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το δικαίωμα στη λύθη, δεδομένου ότι αυτός που συγκέντρωσε τα προσωπικά δεδομένα, είτε είναι στο σελίδα είτε όχι, ε, δεν τα έχει πλέον γιατί τα έχει μεταπολίσει. Οπότε πολύ δύσκολο να επιστρέψει κανείς και να ζητήσει να διαγραφεί από έναν κατάλογο εκ των υστέρων. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι ταυτόχρονα με τον κανονισμό για τη συγκέντρωση αυτών των δεδομένων θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το θέμα της αγοράς, της ανταλλαγής δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί αν δηλαδή θα το επιτρέψουμε, αν θα το απαγορεύσουμε και υπό ποια μορφή. Διότι αυτό που διαφεύγει σε όλους ακόμα και στον, ε, σε αυτόν ο οποίος πρώτος συγκέντρωσε τα στοιχεία είναι τα στοιχεία αυτά. Φυσικά απέναντι σε τρίτες χώρες <laughs> συμφωνώ με την εισηγήτρια και την κυρία Βισταμπεζέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδαμε με το SWIFT ότι το θέμα είναι εξαιρετικά λεπτό. Είναι, και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρξουν κανόνες. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες πρέπει να προστατεύουν τους ευρωπαίους πολίτες. Ακόμα και όταν θα πρέπει να εφαρμόζονται απέναντι σε τρίτους ή ε, σε τρίτες χώρες ή σε παρόχους που βρίσκονται σε τρίτες χώρες και στα κοινωνικά δίκτυα είδαμε ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν ε, περιορίσει την εγκατάσταση κοινωνικών δικτύων επειδή οι... δεν τους ε, θεωρούσαν επαρκή την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Συμφωνώ επίσης με τη Μαρία Λγκαλό που λέει ότι ότι δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στη συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ε, ηλεκτρονικά. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τα χαρτιά και τη συγκέντρωση, τη συλλογή χειρόγραφων. Ε, διαπίστωσα, εγώ ανακάλυψα ότι οι, οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών χρησιμοποιούν τα δεδομένα που κατέχουν, δηλαδή τις διευθύνσεις, τις ταχυδρομικές διευθύνσεις, τις επεξεργάζονται και επίσης τις μεταπολούν. Σε διαφημιστικές εταιρείε που τις χρησιμοποιούν για ταχυδρομική διαφήμιση, δηλαδή σε ένα φάκελο με το όνομα και τη διεύθυνσή σας. Λοιπόν, από τη στιγμή που συγκεντρώνονται ε, ταχυδρομικές διευθύνσεις, γίνεται, δημιουργείται ένα προφίλ ανάλογα με το φύλλο, την περιοχή κατοικία, την ομάδα ε, ηλικίας ηλικία κλπ. Σα δημιουργούν ένα προφίλ και από εκεί και πέρα πολλούνται κατάλογοι προς ε, διαφημιστικές εταιρείες. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να ασχοληθούμε όταν δημόσιοι φορείς ή μη δημόσιοι φορείς και επιχειρήσεις προχωρούν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Θα πρέπει τουλάχιστον να διερωτηθούμε για να δούμε πώς θα παρέμβουμε σε αυτό το σημείο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη η έκθεση αυτή. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο φτάνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπρόσωποι των αρχών προστασίας δεδομένων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην ήθος την ημέρα ε, προστασίας δεδομένων ε, έρχονται όλοι οι εκπρόσωποι και συναντιούνται εδώ στις Βρυξέλλες. Εγώ συναντιούμαι πάρα πολύ συχνά με τον Πολωνό επόπτη της προστασίας των δεδομένων, ο οποίος μου είπε ότι ε, σπανίως ε, υπάρχει μέρημνα για κάποια θέματα σε εθνικό επίπεδο όταν θα έπρεπε ε, να υπάρχουν θέματα προστασίας δεδομένων. Δηλαδή τι εννοώ, ότι σπάνια κάποιο ε, μπορεί να ξεκινήσει να ενεργοποιήσει τον ολόκληρο το μηχανισμό για την προστασία των δεδομένων του. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν ξεκίνησε η συζήτηση για την άκτα, ο Ευρωπαίος Επόπτης ε, Προσωπικών Δεδομένων απέστειλε μια γνωμοδότηση στην πολωνική κυβέρνηση και στη γνωμοδότηση αυτή υπήρχαν ε, κάποιες ε, ε, προτάσεις οι οποίες έγιναν αποδεκτές στην τελευταία ολομέλεια, σύνοδο ολομέλειας εδώ. Ο Πολωνός όμως υπουργό ούτε καν τα διάβασε. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι γίνεται σε κάθε χώρα και ίσως θα έπρεπε και στην έκθεση αυτή να πούμε ότι θα πρέπει να μιλούμε και να συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι επόπτες προσωπικών δεδομένων από όλες τις χώρες μέλη. Όσον αφορά τώρα το δικαίωμα στη διαγραφή των δεδομένων κάποιου. Μπορεί να μην μπορούν να κατανοήσουν όλοι για ποιο λόγο χρειαζόμαστε αυτό το δικαίωμα. Θα είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε τους ε, ε, παρόχους να ξεχάσουν, ε, να διαγράψουν τα δεδομένα και να μας ξεχάσουν. Επομένως, ό,τι και να κάνουμε δεν θα έχει αποτέλεσμα. Τώρα, η πόλη των δεδομένων είναι ένα επιπλέον πρόβλημα, αλλά η διαρροή δεδομένων είναι κάτι το οποίο είναι πλέον πάγια πρακτική. Δείτε, για παράδειγμα, τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες πολύ συχνά δεν φροντίζουν τα δικά μας τα δεδομένα. Μετά από κάποια κραυγαλαία παραδείγματα, διαπιστώσαμε ότι κάποιος ε, μπορεί να βρεθεί, να, να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία του ε, και μάλιστα στοιχεία αρκετά προσωπικά, ε, ασθένειες οι οποίες έχει περάσει ή οτιδήποτε άλλο. Και να μπορεί κάποιος να εξετάσει σελίδε και να διαπιστώσει η ασφαλιστική εταιρεία ότι ο ασφαλισμένος του, για παράδειγμα, ε, πάσχει από AIDS. Πολύ συχνά είναι απαραίτητο να δίνεται η έγκρισή μα για να δημοσιοποιούνται κάποια δεδομένα μα. Για παράδειγμα, όταν αγοράζω κάτι πρέπει να δώσω την συγκατάθεσή μου γιατί αλλιώ δεν έχω δικαίωμα να αγοράσω κάτι. Ορισμένε φορέ δηλαδή δεν έχουμε δικαίωμα επιλογή Για να αγοράσουμε κάτι μέσω διαδικτύου πρέπει να ε, δώσουμε τα στοιχεία μα. Υπάρχουν επίσης επιχειρήσεις οι οποίες είναι, ε, ειδικεύονται ακριβώς στη συλλογή των δεδομένων. θα μπορούσαμε να τις αποκαλέσουμε επιχειρήσεις φάντασμα ή και απλώς παράνομες επιχειρήσεις, διότι πολλές φορές δεν είναι γνωστές. Παραδείγματο χάρη, μου στέλνουν ένα έντυπο και μου λένε ότι μου προσφέρουν κάποιο προϊόν ε, στη τιμή του ενός ή των δύο ευρώ. Στην πραγματικότητα βέβαια δεν είναι τόσο σημαντική η αγορά του προϊόντος, αλλά ε, η συμπλήρωση του εντύπου, γιατί η επιχείρηση που ασχολείται με τα θέματα αυτά ενδιαφέρεται να λάβει τα στοιχεία μας και κατόπιν να μεταπολεμήσει τα μεταπολίσει σε κάποιον άλλον. Υπάρχουν δηλαδή μία σειρά από επιχειρήσεις φάντασμα οι οποίες στην πραγματικότητα ούτε πουλούν προϊόντα ή αγαθά και υπηρεσίες αλλά ε, χρησιμοποιούν τα στοιχεία του που του δίνουμε για να τα μεταπολίσουν σε άλλους. Η συνάδελφο Γκαλό έχει μεγάλη πείρα στον τομέα αυτό και ε, φυσικά μας ε, περιμένει πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Η κυρία Τάιν. Ευχαριστώ. Πολύ να θα θέλω να κάνω μια παρατήρηση στο όσο κυρία Για την ε, προϋπόθεση να υπάρχει μια επιπτεύουσα αρχή και ότι δεν θα πρέπει να συνδέεται η προστασία των δεδομένων με τον ε, αριθμό, η επιλογή μάλλον ε, της επιχειρήσης στους μικρομεσαίες με τον αριθμό μόνο. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε με, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα. Γιατί υπάρχει παραδείγματι τώρα κάτι στις υπηρεσίες μας που δεν είχαμε παλιά, έναν αρμόδιο για την ασφάλεια παραδείγματι. Η ε, εξέλιξη αυτή ξεκίνησε μετά την 11η Σεπτεμβρίου και μια ολόκληρη διαδικασία με τη σχετική οδηγία που ξεκίνησε μετά από αυτήν ε, την ε, τραγωδία. Άρα Υπάρχουν ε, σε επίπεδο ακόμη και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, ε, αρμόδιοι, επιφορτισμένοι με θέματα ασφάλειας, με θέματα εργονομίας, εκείνο το άλλο, που πάντοτε βέβαια συνεπάγονται και επιπλέον κόστος. Φυσικά δεν έχει κανένα νόημα να θεσπίσουμε την αρχή του υπεύθυνου ασφάλεια προσωπικών δεδομένων αν δεν είναι ικανό, αν δεν έχει τι γνώσει δηλαδή να επιτελέσει το έργο αυτό αποτελεσματικά. Άλλωστε το έχουμε δει και στη Γερμανία ότι πολύ συχνά δεν λειτουργεί ε, το σύστημα αν δεν υπάρχει κατάλληλη εξειδίκευση. Αλλά α μην θεωρούμε περιττό το να αναλάβει κάποιος από τους ε, εργαζομένους μιας επιχείρησης αυτό το καθήκον μπορεί να ανατεθεί και σε εξωτερική αρχή η επιχείρηση. Μπορεί να υπάρξουν επιχειρήσεις οι οποίες θα εξειδικευτούν σε αυτό, αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ότι ειδικά αν πρόκειται για υπερσυνοριακή αρμοδιότητα ε, θα είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα. Κύριο Σιέφκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση αποδεικνύει πόσο μεγάλη σημασία δίνουμε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχω μια παρατήρηση. Εγώ διαφωνώ με τη Λίντια και τα επιχειρηματά της. Δηλαδή, ότι η άκτα μας απέδειξε ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Δεδομένων είναι άχρηστος γιατί η πολιτική κυβέρνηση δεν τον άκουσε. Είπαμε ότι ε, μπορεί να συμβούν κάποια πράγματα πέραν της άκτα. Η άκτα βέβαια μου φέρνει στο νου κάτι άλλο. Γιατί κινητοποιηθήκαμε όλοι και μας συγκίνησε τόσο πολύ το θέμα της άκτα. πότε χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μας, ε, για παράδειγμα, για να δημιουργήσουμε το προφίλ ε, κάποιου. Στην πραγματικότητα, ε, το πιο συχνό φαινόμενο κλοπής προσωπικών δεδομένων είναι μέσω του διαδικτύου. Και τη σήμερα ημέρα βρισκόμαστε υποχρεωμένοι να περιορίσουμε την ελευθερία του διαδικτύου, ώστε να υπάρχει προστασία των προσωπικών μας δεδομένων. Ούτως ή άλλως αυτή η ελευθερία δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο διαδίκτυο είτε πρόκειται για κλοπή προσωπικής ταυτότητας, είτε πρόκειται για κλοπή προσωπικών δεδομένων, ε, τα δύο θέματα είναι αλληλένδετα. Ε, και εμείς από τη μια λέμε ναι και από την άλλη λέμε όχι. Αν ασχοληθούμε λοιπόν με όλο το πακέτο που αφορά και τα προσωπικά δεδομένα και την ε, πνευματική ιδιοκτησία, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα στοιχεία και αυτή είναι η έκκληση που σας κάνω. Δεν θα πρέπει να χαθούμε στις λεπτομέρειες και να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να πούμε ότι είμαστε δυσαρεστημένοι, διότι ε, θα βρεθούμε ενώπιον της ίδιας ιστορίας. Jetzt dazu veranlasst mich äh, äh, auch noch zu Wort zu melden. Äh, η κυρία Τάουν ε, θα λάβει βεβαίω και εκείνη το λόγο. Θα ήθελα να πω όμω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσει οι οποίε έχουν εργαζομένους με μεγαλύτερη προστασία προσωπικών δεδομένων από ό,τι κάποιοι άλλοι. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί να υπάρχει μια επιχείρηση η οποία κάνει επεξεργασία μόνο και έτσι μπορεί να έχει λίγους εργαζομένους αλλά μεγάλο αριθμό πελατών, μεγάλη δηλαδή επικοινωνία με κοινό και άρα έχει εκεί στο θέμα του πελατολογίου τη ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα ήθελα δεν να πω εγώ για την ε, πατρίδα μου την Αυστρία ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο εργοδότης απαιτεί από τον εργοζόμενο να ε, υπογράψει μία σύμβαση προστασίας των δεδομένων και για να μην μπερδεύονται τα πράγματα θα ήθελα να πω ότι βεβαίως δεν πρέπει να επιβληθούν περί να επιβληθεί περί τη γραφειοκρατική επιβάρυνση, φόρτος, αλλά από την άλλη ο εργαζόμενος σε μια μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να μετατραπεί σε έναν ε, πολίτη δεύτερης κατηγορίας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. συγγήτρια, κυρία Γκαλό, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ομολογώ ότι χαίρομαι με την αντίδραση των συναδέλφων διαπιστώσω, διαπιστώνω ότι αυτό το θέμα του ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από το δικαίωμα των δικαιωμάτων παρακολούθησης. Χαίρομαι. Και πρέπει να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την Εύα ότι ότι παραδείγματο χάρη στην περίπτωση του cloud computing θα πρέπει οπωσδήποτε να αναπτύξουμε κέντρα δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλάβουν την εξυπηρέτηση, να προσφέρουν την υπηρεσία του cloud. Δεν μπορεί επάπειρο να εξαρτώμαστε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω επίσης να ε, καθησυχάσω τη Φρανσουάς Καστέξ που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα για την ε, νομοθετική πρόταση της οποίας το κεφάλαιο 4 ασχολείται με την ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας. Αναφέρεται σε κοινή ευθύνη και υπάρχει και η ευθύνη του υπεργολάβου. Δηλαδή, σε αυτό το κεφάλαιο 4, αν δεν είμαστε απολύτως ε, ε, ικανοποιημένοι, μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, αλλά θεωρώ ότι είναι αντίστοιχο και έχει αρκετές ενδιαφέρουσες ιδέες. Όσον αφορά τα τρίτα κράτη και τη μετάδοση, μεταφορά δεδομένων, αυτό που είπε η Εύα Λίχτεμπεργκ εξακολουθεί να ισχύει. Δεν μπορούμε να, πάρουμε να δώσουμε υπερβολικά μεγάλη πρωτοβουλία σε κάθε κράτος μέλος. Θα πρέπει να καταλήξουμε στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εναρμόνιση. Παρότι είμαι πολύ παλιά βουλευτής, γνωρίζω πλέον ότι υπάρχουν και όρια σε αυτή την εναρμόνιση. Όλοι ονειρευόμαστε, αλλά όταν αρχίζουμε τη συζήτηση ενός κειμένου και καταλήγουμε σε συνένεση, <laughs> διαπιστώνουμε ότι πολύ συχνά υπάρχει ένα όριο πάνω από το οποίο δεν μπορούμε να περάσουμε. Ένα όρατο όριο πάνω από το οποίο δεν μπορούμε να περάσουμε. Νομίζω ότι το θέμα αυτό μπορεί να μας απασχολήσει ε, για υπέρ του γενικού συμφέροντος όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας από μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορούμε να κλείσουμε αυτό το θέμα σήμερα στη διάταξη. Και πάμε, μια και δεν έχουμε εδώ ακόμα την κυρία Μακάρθη, στον κύριο Καρύμ. Τα σημεία 8 και 9. Μια στον παρουσίαση. Και μετά την παρουσίαση για το Impact Assessment. Το δεν ξέρω αν είναι εδώ. Μάλιστα. Ναι, είναι εδώ. Επομένω, ο κύριο Καρή μα λέει πρώτο το λόγο. Chairman, thank you. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ. Έχω μια αρκετά μακροσκαλή παρουσίαση να κάνω στην Επιτροπή σήμερα. Έχοντας όμως κατά νου και τη φύση του θέματος με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, ε, ελπίζω να δείξουν κατανόηση οι συνάδελφοι, διότι πρέπει να επισέλθω σε κάποιες λεπτομέρειες. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία. Ο κ. Μασί Πιντάλγο είναι εδώ, ε, αλλά και άλλοι συνάδελφοι υπήρξαν ιδιαίτερα συνεργάσιμοι ε, όταν τους τηλεφωνούσα για να μου δώσουν τις απόψεις τους, αλλά φυσικά και την εμπειρογνωμοσύνη τους. δράτω με τις ευκαιρίες της παρουσίασης του εγγράφου εργασίας που ουσιαστικά είναι άλλο ένα τμήμα στη διαδικασία της μεταρρύθμισης και επανεξέτασης ε, της διαδικασίας ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ συνειδητοποίησα ότι ανεξάρτητα από τις ε, διστάμενες απόψεις που μπορεί να είχαμε μεταξύ των συναδέλφων της Επιτροπής, υπάρχει ε, ένας κοινός στόχος και αυτός είναι να παρουσιάσουμε ε, μία δέσμη προτάσεων που θα ενισχύσουν τους Ευρωπαίους πολίτες και θα βελτιώσουν την ποιότητα των ελέγχων που γίνεται ε, και φυσικά θα βοηθήσουν και τις επιχειρήσεις. Το έγγραφο εργασία θα πρέπει από πλευρά μου τουλάχιστον ε, να το θεωρήσετε ως έγγραφο συζήτησης που αφορά κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Πολλά από αυτά τα θέματα είναι γνωστά σε όσους παρακολουθούν τη συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις στην ε, ε, πολιτική ελέγχων, αλλά υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε εξίσου, εξίσου και αυτή τη στιγμή δεν έχουν λάβει τη δέουσα προσοχή όπως για παράδειγμα την ανάγκη να βελτιωθούν οι εκθέσεις ε, ελέγχων, να εξετάσουμε το ρόλο των επαγγελματικών φορέων και την θέσπιση διεθνών προτύπων ε, για τους ελέγχους αυτούς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Γενική Διεύθυνση που μου έκανε μια εκτίμηση της αξιολόγησης αντικτύπου που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η πρώτη τέτοια εκτίμηση που ετοιμάζει ε, για την Επιτροπή μας και ελπίζω κύριε Πρόεδρε να μην είναι και η τελευταία. Πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο έγγραφο το οποίο θα μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε την άποψή μας και στην Επιτροπή μας εδώ αλλά και σε όλο το Κοινοβούλιο. Και πρόκειται και ένα έγγραφο το οποίο παρουσιάζει κάποιες σημαντικές ανησυχίες και θα ήθελα να ακούσω και την ε, άποψη της Γενικής Διεύθυνσης αργότερα εδώ συνεδρίαση. Όσον αφορά τώρα την προσέγγισή μας για το θέμα αυτό, καταρχάς να πω ότι ε, προς το παρόν είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Δεν έχω λάβει κάποια οριστική απόφαση, αλλά η φιλοσοφία που διέπει όλα όσα έχω λάβει κατά νου ε, βασίζεται σε δύο στοιχεία. Να ενισχύσουμε την ποιότητα των ελέγχων και να υπάρχουν καλύτερες πληροφορίες για τους ε, ελεγκτές. Ε, υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία όμως δεν με αποσχολούν τόσο ε, σημαντικά. Ε, δεν ε, επαφίεται στους νομοθέτες να καθορίσουν το αριθμιστικό πλαίσιο. Αυτό είναι αρμοδιότητα της αγοράς και των αρχών ανταγωνισμού. Αυτό βέβαια κύριε Πρόεδρε δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση έχει σχέση και επιπτώσει στην αγορά δεν θα τη λάβουμε υπόψη. Ε, θα πρέπει να δούμε και ε, πώς θα ισοσκελίσουμε τα διάφορα στοιχεία. Ποια είναι λοιπόν τα θέματα που μας αποσχολούν. Θα προσπαθήσω να σας τα απαριθμίσω τα θέματα που έχουμε στο έγγραφο εργασία και στη συνέχεια θα αναφερθώ σε πιο συγκεκριμένα σημεία τα οποία έθιξε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο προτάσεων ε, το οποίο θα πρέπει να λάβει υπόψη ε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς, όσον αφορά τη δομή της αγοράς και την ανεξαρτησία της. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για υποχρεωτική εκπεριτροπής ε, διαδικασία ελέγχων. Άκουσα και πολλούς ε, να λένε ότι υπάρχει δυνατότητα να έχουμε κοινούς ελέγχους, να υπάρχουν ε, υποχρεωτική έλεγχη. Ε, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα για την εξαιρετική ε, εξωτερική εκπεριτροπή διαδικασία ελέγχων και έχω κάποιες απόψεις στο έγγραφο εργασίας. Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις οι οποίες θεωρώ ότι είναι υπερβολικές. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα αυξημένης ποιότητας σε πεδίο δεκαετίας το οποίο ίσως είναι δυνατόν να επιτύχουμε αλλά δεν είναι δυνατόν να βελτιώσουμε την ποιότητα ευθύ εξ αρχής. οι νέοι ελεγκτείς είναι υποχρεωμένοι να μάθουν και να αμφισβητούν τις πρακτικές ε, μιας επιχείρησης ε, στις τελικές τους εκθέσεις. Ε, και αυτό ίσως να θεωρηθεί ότι έξι χρόνια είναι μικρό διάστημα για να υπάρχει αυτή όσο εκπεριτροπής έλεγχος και μπορεί να δημιουργηθούν και ερωτηματικά για την ε, βάση ε, της πρότασης. Εμείς ως Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικό πώς θα επηρεάσει αυτή, ε, ε, η πρόταση την αγορά, διότι υπάρχουν και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Επίσης υπάρχουν και κίνητρα ίσως για κοινού ελέγχου, ε, τα οποία όμως είναι αμφισβητήσιμα, κυρίως λόγω του κόστους που μπορεί να βασίζεται από την εμπειρία, από τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι έλεγχοι σε κάθε κράτος μέλος ε, και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και ε, σαφή προβλήματα επανάληψης των ίδιων εργασιών, ε, κατάλληλης πολιτικής ε, και ορισμένα φορές δεν υπάρχουν και αρκετές ενδείξεις ότι έχει βελτιωθεί η ποιότητα. Εγώ κύριε Πρόεδρε δεν είμαι πεπισμένος ότι τα αρνητικά μπορούν να ισοσταθμιστούν από τα θετικά στοιχεία και ότι η παρέμβαση με ρυθμιστικά μέσα μπορεί να μας βοηθήσει. Οι κοινοί έλεγχοι φυσικά υπάρχουν ως έννοια και ορισμένες φορές ε, μόνο ένα μικρό ποσοστό μπορεί να είναι κοινό ε, για τον έλεγχο σε μια ελεγκτική διαδικασία. Λαμβάνονται υπόψη και τα ωφέλη και της ε, ανεξαρτησίας για την ποιότητα, η οποία δεν είναι ίσως τα ίδια, συγγνώμη, τα ωφέλη δεν είναι τα ίδια όταν έχουμε κοινούς ελέγχους. Τώρα, έχει συζητηθεί επίσης και το θέμα του ε, να γίνεται υποχρεωτικά ε, νέα προσφορά ε, αλλά φυσικά όταν υπάρχουν νέε μειοδοτικέ διαδικασίε υπάρχει επιπλέον κόστο, ιδίω όταν συμμετέχουν μικρομεσαίες επιχειρήσει, οι οποίε θα πρέπει να επιβαρυνθούν με αυτό το επιπλέον κόστο και θα πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες ε, ε, γίνεται μια νέα διαδικασία μειοδοτικού διαγωνισμού χωρίς να υπάρχει προστιθέμενη αξία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, έχουμε τη δυνατότητα νέου μειοδοτικού διαγωνισμού σε επίπεδο δεκαετίας. Ίσως το χρονικό διάστημα να μην είναι το σωστό, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι ο καλύτερος τρόπος να μετριάσουμε ε, την κατάσταση και να μην έχουμε υπερβολικό κόστος και για όσους καταθέτουν προσφορές, αλλά και για τις δημόσιες αρχές και να μην επιβαρύνουμε σημαντικά τους μειοδετικούς διαγωνισμούς. Υπάρχουν και κάποια προβλήματα που αφορούν τη δομή της αγοράς ε, και προκύπτουν από το γεγονός ότι δεν είναι παντού με τον ίδιο τρόπο δομημένη η αγορά και θα πρέπει ε, να δούμε κάποια προβλήματα που προκύπτουν από εκεί και δεν είναι προφανή. Θα πρέπει να έχουμε μια νέα προσέγγιση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιωτερότητες και των εθνικών αργορών και των εμπορικών προσφορών ακόμα και ε, σε ε, υποκατηγορίες των αγορών οι οποίες θα μπορούσαν να ε, αντιμετωπίσουν προβλήματα. Όσον αφορά τώρα τις εκθέσεις για τους ελέγχους λόγω των αλλαχών που μπορούμε να κάνουμε, ε, οι εκθέσεις μπορεί να είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία της μεταρρύθμισης. Από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, διαπιστώνω ότι εξετάζουν πολύ το ζήτημα αυτό και εξετάζεται και στα πλαίσια του IIASP και θα πρέπει να διαβεβαιωθούμε ότι οι τελικές μας προτάσεις θα λάβουν υπόψη τους και τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές αν θέλουμε να έχουμε τον ηγετικό ρόλο διεθνώς, θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση που θα οδηγεί ε, ε, σε καλά αποτελέσματα για τον τελικό πελάτη του ελέγχου, τους μετόχους και τους επενδυτές. Θα πρέπει να έχουμε μια διαδικασία όπου θα έχουμε ένα κατάλογο και θα ελέγχουμε ότι έχουν επιτευχθεί τα στοιχεία όλα, ε, αλλά χωρίς να χάνουμε και από το επιπρόσθετο όφελος που μπορούμε να έχουμε. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την αρχή less is more, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το λιγότερο θα πρέπει να βασίζεται στην ποιότητα. Ε, και ίσως να, ε, αν δεν προσέξουμε, να οδηγήσουμε σε ελέγχους οι οποίοι θα γίνονται βεβαιασμένα και δεν θα βελτιώσουμε την ποιότητα. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις εκθέσεις λοιπόν και θα σας ε, προτείνω και κάποια στοιχεία στον τομέα αυτό εν ευθέτω χρόνο. Τώρα, η Επιτροπή Ελέγχου. Ένα βασικό στοιχείο για να βελτιώσουμε την ποιότητα ενός ελέγχου είναι να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε αποτελεσματική και ενεργό συμμετοχή των Επιτροπών Ελέγχου. Οι Επιτροπές Ελέγχου θα πρέπει ε, να είναι τμήμα της γενικότερης δέσμευσης για καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση και θα πρέπει να φροντίσουμε ότι στηρίζουμε παρκώς αυτές τις δομές. Είναι ε, ανάμεικτες οι εμπειρίες που έχουμε στα κράτη-μέλη και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια βελτίωση και ενίσχυσή των. Η Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον διορισμό και στην εποπτεία της διαδικασίας ελέγχου και θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά την εντολή τους όταν θα περάσουμε στα σημεία αυτά. Παραδείγματο χάρη, ε, η δυνατότητα να γίνονται αποδεκτές, ε, να προσφέρονται αποδεκτές υπηρεσίες που δεν έχουν σχέση με τον έλεγχο και θα πρέπει να γίνεται κατάλληλος διαχωρισμός μεταξύ του ελεγκτή και της διαχείρισης της επιχείρησης και ε, να παρέχουμε και να φροντίσουμε να αποφεύγουμε σύγκρουση συμφορώντων. Επίσης υπάρχει ανάγκη να σκεφτούμε τρόπους ώστε η Επιτροπή Ελέγχου να συμμετέχει με τους επενδυτές, να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία και να μπορούν οι επενδυτές ε, να εμπλακούν στην όλη διαδικασία. Και επίσης κύριε Πρόεδρε, ε, στοιχεία για τα θέματα της εμπιστευτικότητας μπορεί να είναι πολύ σημαντικά για τα βασικά προβλήματα ελέγχων που μπορεί να ανακύψουν στη διάρκεια του ελέγχου. Η εμπιστευτικότητα βέβαια έχει και κάποια όρια για το τι πρέπει να αποκαλύπτεται ε, και δεν θα πρέπει να ε, υποχρεούνται οι ελεγκτές και η Επιτροπή Ελέγχου ε, να κάνουν τις συζητήσεις τους υπογείως. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις βελτιώσεις στον τομέα αυτό. Τώρα κύριε Πρόεδρε, οι υπηρεσίες που δεν είναι ελεγκτικού χαρακτήρα. Μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη μπορούσαν να καθορίσουν το δικό τους καθεστώς για το τι γίνεται για τις ε, υπηρεσίες ε, ε, που παρέχονται από ελεγχτές αλλά δεν είναι ελεγκτικές υπηρεσίες. Αυτό ε, με οδήγησε σε μία εξέταση να δω τι γίνεται σε κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά. Όπω σα είπα προηγουμένω, θεωρώ ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα μπορούσε να συμμετέχει στι διαδικασίε όταν υπάρχει ένα κατάλογο ε, καθορισμένων υπηρεσιών που θα μπορούσαν να προσφέρονται, ε, αλλά θα πρέπει να ε, μπορούμε να το κάνουμε με ικανοποιητικό τρόπο. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτής της γκρίζας λίστας και ενώ ενός ε, διεθνούς φορέα όπως είναι το δικαστήριο ESPA και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση από αυτού. Όσον αφορά τώρα τις ε, ελεγκτικές υπηρεσίες, θεωρώ εδώ ότι η πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ε, για τη σύγκρουση συμφορώντων όταν δεν παρέχονται υπηρεσίες, ε, ε, όταν παρέχονται συγγνώμη, υπηρεσίες που δεν είναι ελεκτικές και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι γίνεται. Δεν μπορεί οι ελεγκτές να είναι υποχρεωμένοι να παρετηθούν ή να πρέπει να λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένο όριο για να μην ε, γίνει διαχωρισμός μεταξύ ελεγκτικών και μη ελεγκτικών υπηρεσιών. Και φυσικά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή η πρόταση. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, εφαρμογή διεθνών προτύπων σε γενικές γραμμές υπάρχει συμφωνία ότι η εφαρμογή του ISIS θα ήταν προς όφελος όλων. Θα μας βοηθήσει να έχουμε ένα κατάλληλο βαθμό εναρμόνισης, θα μας επιτρέπει να έχουμε μεταφορά από το ένα στο άλλο και θα έχουμε και μια βάση σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων εκθέσεων. Ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία βέβαια τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε για να δούμε αν θα μπορούσαμε να έχουμε το ISA συν και όχι το ISA πλην. Ε, καταρχάς, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη απόκληση μεταξύ των υπηρεσιών που ε, προσφέρονται και ε, θέλουμε όμως να έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε και σύγκριση μεταξύ λογιστικών προτύπων, οπότε χρειάζεται και κατάλληλη ευελιξία. Τώρα, μία πτυχή που δεν αναφέρεται συχνά είναι ο ρόλος επαγγελματικών φορέων στην εξέλιξη του ελεγκτή δεν με πείθει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ε, θα ακυρώσει πολλές από αυτές τις δραστηριότητες αυτών των φορέων και θα υποχρεώνει τις εθνικές αρχές ε, να κάνουν πολλά από τα όσα κάνουν αυτοί οι φορείς. Εγώ θεωρώ ότι καλό θα ήταν να αποφασίσει το κάθε κράτος μέλος ανάλογα με τις διαφορές που υπάρχουν στις πρακτικές τους και τις δυνατότητες που έχουν τι θα πρέπει να γίνει. Η συζήτηση τώρα ε, για το κατά πόσον θα πρέπει να έχουμε κανονισμό ή οδηγία είναι πολύ σημαντική, αλλά μας οδηγεί στη γενική παρατήρηση την οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Κατά πόσον το καλύτερο μέσο για να επιτύχουμε πολλούς από αυτούς τους στόχους πολιτικής είναι ο κανονισμός, όταν τα περισσότερα από αυτά που προτείνονται θα μας επηρεάσουν ε, σε διαφορετικό επίπεδο, ανάλογα με την κατάσταση σε κάθε χώρα αιτιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιεί κανονισμό είναι πολύ γενικόλογη και δεν μας εξηγεί ε, για κάποια στοιχεία τα οποία είναι ετερογενή όσον αφορά τους ελέγχους σε κάθε κράτος μέλος. Ίσως θα ήταν πιο σωστό να υπάρχει μια οδηγία και η Επιτροπή μας θα έπρεπε να εξετάσει μήπω αυτή είναι η καλύτερη προσέγγιση και όχι ο κανονισμός. Εμείς λοιπόν ως Κοινοβούλιο Ω προ τη διαδικασία, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να λάβουμε υπόψη ε, τι γίνεται ε, και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, διότι μέχρι τούδε είμαστε μάλλον αρκετά ελαστικοί. Ε, υπάρχει η... Ε, διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο της Επιτροπής Ανταγωνισμού που κάνει μια ίδια διαδικασία έρευνας, αλλά δεν νομίζω ότι αρκεί μόνο αυτή. Θα μπορούσαμε να δούμε και τι κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε στο BCLB για την ανεξαρτησία των ελεγκτικών φορέων και να λάβουμε υπόψη και άλλα θέματα εξωτερικού συστήματος εκπεριτροπής. Ε, διάβασα κάπου πρόσφατα ότι το σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο βρετανικός τρόπος για να απορρίψουμε τις μεταρρυθμίσεις. Δεν συμφωνώ. Ε, υπάρχουν κάποιες απαιτήσει και καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη μεταρρύθμισης. Κύριε Πρόεδρε, σας έχω πει και στο παρελθόν ότι δεν είναι εναλλακτική λύση το να παραμείνουμε ε, στο καθεστώς που έχουμε και τώρα. Και το επαναλαμβάνω ότι ε, η προσέγγιση μου είναι ακριβώς ότι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα. Η διαδικασία όπως έχει αυτή τη στιγμή κύριε Πρόεδρε είναι η εξή. Υπάρχει ένα σχέδιο έκθεσης το οποίο θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο αρχές Οκτωβρίου η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, ε, ψηφοφορία αρχές Δεκεμβρίου. Και αυτό το χρονοδιάγραμμα συνάδει και με την προσέγγιση που έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει η Κυπριακή Προεδρία. Οι συνάδελφοι που ήταν εδώ το πρωί άκουσαν ε, ε, ότι έθεσα και σχετική ερώτηση στον Υπουργό που μίλησε στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Μάσεπ, Budu, Lichtenberger, Time. Και θα, θα ακούσουμε και την ε, Διεύθυνση για την Αξιολόγηση Επιπτώσεων. Ε, παρακαλώ. Ο κύριος Ντάλγο. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον φίλο Καρύμ. Νομίζω ότι αυτό που είπατε, η σημασία της ποιότητας του ελέγχου και το πόσο σημαντικό είναι οι τελικοί χρήστες, είτε είναι μέτοχοι είτε επενδυτές, είναι αυτή που θα πρέπει να λαμβάνουμε κυρίως υπόψη ε, στον τρόπο με τον οποίο θεωρούμε το πρόβλημα μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους και μάλιστα όχι μόνο συμφωνώ αλλά θα είμαι ένθερμος υποστηρικτής σε αυτό και κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει σύμπτωση απόψεων. Εκεί όμως που προκύπτει ένα σημαντικό πρόβλημα είναι όταν ο εισηγητής μας λέει ότι δεν θα προσπαθήσουμε να παρέμβουμε στην διαχείριση της αγοράς. Εμείς δεν θέλουμε να παρέμβουμε στη διαχείριση της αγοράς. Η αγορά αυτή τη στιγμή αποτελεί αντικείμενο χειραγώγησης. Και απόλυτης χειραγώγησης. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε κατεπηγόντως οδηγό, οδηγία τώρα εν καιρό κρίσης. Είναι τεράστια χειραγώγηση της αγοράς και μάλιστα σε τέτοιο σημείο που είμαι βέβαιος ότι από, κάποιοι από αυτούς που βρίσκονται εδώ ε, και παρακολουθούν τη συζήτηση εκπροσωπεί μία από τις τέσσερις μεγάλες επιχειρήσεις ε, που χειραγωγούν την αγορά, τους Big Four. Και είμαι βέβαιο. βέβαια δεν μπορεί να έρθει κανείς εδώ να μας ομολογήσει, αλλά ε, υπάρχουν αυτοί οι big four οι οποίοι χειραγωγούν την αγορά και εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια όταν γίνεται κάτι τέτοιο. Επιπλέον, οι χειρότερες ε, προβλήψεις μου για τις νέες αυτές μελέτες ε, αντικτύπου επιβεβαιώθηκαν διότι σήμερα μαζί με τις νέες προτάσεις ε, του εισηγητή ε, έχουμε και ακριβώς αυτά τα ίδια στοιχεία. Περιέργως, όπως τα έλεγαν οι στατιστικοί, υπάρχει μία ε, αντιστοιχία μεταξύ αυτών των τεσσάρων εγγράφων, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να έχουν γίνει το καθένα ανεξάρτητα από το άλλο. Στη μελέτη αντικτύπου του Κοινοβουλίου νομίζω ότι έχουμε το πιο ε, καλό όνειρο θερινής νυχτής ε, ε, της Βρετανίας. Όνειρο θερινής νυχτός θα έλεγε ο Σέξπιρ. Ή ήταν όνειρο θερινής νυχτός με ελληνική μυθολογία αυτό το οποίο μας παρουσίασε. και θα χρησιμοποιηθεί και ως όπλο για να εμποδίσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ε, υπάρχει και μία μελέτη αντικτύπου που βασίζεται στη μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ακόμα χειρότερα. Δεν έχουμε εδώ κανένα στατιστικό στοιχείο και κανένα επίσημο στοιχείο. Πρόκειται για μια μελέτη η οποία έχει ένα σαφή πολιτικό ε, προσανατολισμό και λέει ότι το γεγονός ότι υπάρχουν ε, μεγάλα προβλήματα στην αγορά δεν είναι πρόβλημα αυτό καθ' αυτή. Αυτό το έχω ακούσει και πριν ξεκινήσει η συζήτηση εδώ και πριν κάνουμε τις ακροάσεις που κάναμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ακούσουμε τους εκπροσώπους ε, της Royal Bank of Scotland. Το ίδιο ακριβώς πράγμα μας είχε πει και ο εκπρόσωπος της Royal Bank of Scotland όταν ήρθε. Ουσιαστικά πρόκειται για εγκόμιο των μονοπωλίων παγκοσμίω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολιτικό όργανο το οποίο πρέπει να παρουσιάζει πολιτικές προτάσεις και δεν θα πρέπει ε, να αφήνουμε μια γενική διεύθυνση του Κοινοβουλίου να κάνει μια υποτιθέμενη εντός εισαγωγικών ε, ανεξάρτητη αξιολόγηση αντικτύπου. Και ουσιαστικά τι κάνουμε, ε, παρουσιάζουμε ως αμεροληψία τις πολιτικές επιλογές μιας συγκεκριμένη πολιτικής ομάδας. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θεωρώ ότι από μόνο του το μονοπόλιο είναι ε, στρεβλό, υπάρχει ολιγοπόλιο και εγώ είμαι υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν δεσμεύει η πολιτική μας απόφαση αξιολόγηση αντικτύπου. Έχουμε το ελεύθερο να αποφασίσουμε όπως ε, θεωρούμε. Δεν μας δεσμεύει κανείς. Ο συνάδελφος Da, mulțumesc, domnule președinte. Am citit documentul de lucru pregătit de... Κύριε Πρόεδρε, μελέτησα το έγγραφο εργασίας τα θέματα που, έχουμε, που τίθενται εδώ πρέπει να πω ότι είναι πολύ σωστά γιατί ο εισηγητής θέτει κάποια ερωτήματα σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δίνει και κάποιες απαντήσεις. Συνολικά θεωρούμε ότι εμείς, ελπίζω ότι εμείς οι εισηγητές θα μπορέσουμε να απαντήσουμε όλα τα ερωτήματα του βασικού εισηγητή που περιλαμβάνονται στο έγγραφο εργασίας. Θέλω να σας πω και κάποιες προσωπικές απόψεις για το περιεχόμενο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συζητήθηκε με πολλούς συναδέλφους του ΕΛΚ, αλλά και όχι μόνο του ΕΛΚ. Καταρχήν, Δεν θέλω να ξεκινήσω από την μελέτη αντικτύπου που πρόσφατα μας παρουσιάστηκε. Ο συνάδελφος, ο συνάδελφος μας είπε, μίλησε και αυτός για αυτή τη μελέτη. Χαίρομαι για κάτι και το έχω πει και από την αρχή, το οποίο επιβεβαιώνει και η μελέτη. Δεν είναι πολιτική θέση αυτή. Επειδή όμως συμφωνώ με αυτή τη θέση, ίσως εγώ να είμαι υποκειμενικός και να ισχύει, και, ισχύει βέβαια και το αντίστροφο. Πάση περιπτώσει η μελέτη αυτή και διαβάζω αγγλικά. Η συγκεκριμένα η τυχαία ε, σχέση ανάμεσα στο ονομαζόμενο πρόβλημα επιτε, αποτελεσματικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης δεν έχει δειχθεί. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η πρόταση της Κομισιόν στην πρώτο εδάφιο στηρίζεται στην υπόθεση ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ποιότητα των ελέγχων και την ε, κρίση. Εδώ η μελέτη δείχνει το ακριβώς αντίθετο. Άρα, το λέει και η μελέτη, το επιβεβαιώνω και εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα που να αφορά την ποιότητα της υπηρεσίας, αλλά υπάρχει πρόβλημα λόγω της συγκέντρωσης της αγοράς στα χέρια τεσσάρων εταιριών. Ένα πρόβλημα που βεβαίως πρέπει να μελετηθεί, όχι όμως με τον τρόπο που το έκανε η Κομισιόν. Η μελέτη επικρίνει τη λύση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα της συγκέντρωσης των υπηρεσιών στα χέρια τεσσάρων εταιριών. Θέλω να κάνω μία πρόταση στον εισηγητή. Θέλω να δείξω μια, ότι η πρόταση αυτή είναι πολύ καλά μελετημένη. Και θα ήθελα πολύ οι σοσιαλιστές και πράσινοι συνάδελφοι να την δεχτούν θετικά. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό το λιγοπόλιο, αυτές οι τέσσερις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να σπάσει με δύο τρόπο. Δηλαδή να τις χωρίσουμε σε δύο, σε επιχειρήσεις ε, ελέγχου και σε επιχειρήσεις που δεν κάνουν έλεγχο. Πιστεύω ότι σιγά σιγά πρέπει να δοθεί περισσότερος χώρος σε υπηρεσίες που να μην είναι υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου αλλά συμβούλων, Δηλαδή να δώσουμε χώρο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολύ συχνά δίνουν πολύ καλές επιχειρηματικές λύσεις ε, για τις μεγάλες, τις μεγάλες εταιρείες, αλλά που δεν έχουν τη δυνα, διοικητική δυνατότητα να προσφέρουν ε, λύσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο στις μεγάλες επιχειρήσεις, να προσφέρουν υπηρεσίες που να μην είναι υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου και από τη στιγμή που θα αποκτήσουν κάποια αρκετά ισχυρή θέση σε αυτό το χώρο να θεωρηθούν, να λαμβάνουν υπόψη ως επιχειρήσεις παροχής οικονομικού ελέγχου στις μεγάλες επιχειρήσεις. Μπορούμε να θέσουμε ανώτατο όριο στις ε, αμοιβέ των επιχειρήσεων, των ε, οικονομικού ελέγχου και σε αυτές που θα καταβάλουν οι τρίτες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις οικονομικού ελέγχου. Θα είναι μια βαθ... Ε, ε, ένα κλιμακωτό τιμολόγιο αν θέλετε και από εκεί και πέρα θα μπορεί να κάνει την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε θα υπάρχει θέση για τις μικρές επιχειρήσεις και ελπίζουμε ότι αυτές οι μικρές επιχειρήσεις με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να μεγαλώσουν και να γίνουν σημαντικοί παράγοντες στην αγορά αυτή που αργότερα ενδεχομένως θα λαμβάνονται υπόψη, θα τις χρησιμοποιούν οι μεγάλες επιχειρήσεις για να τους παρέχουν ε, υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου και όχι μόνο υπηρεσίες που δεν θα είναι άλλες εκτός από οικονομικού ελέγχου. Θέλω να πω στον εισήγητη, όπως έλεγα και πριν. Δεν θα πρέπει να σπάσουμε στα δύο τις επιχειρήσεις αυτές. Δεν θα πρέπει να δεχτούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να έχουμε επιχειρήσεις λεγόμενες οικονομικού ελέγχου και άλλες χρηματοοικονομικές. Θεωρώ επίσης ότι η υποχρεωτική ανανέωση των συμβολέων ελέγχου δεν είναι η επιθυμητή λύση σε αυτό το λιγοπόλιο αυτό απλώς θα αυξήσει το κόστος για τις επιχειρήσεις. Γιατί αν μια επιχείρηση είναι ικανοποιημένη από τον οικονομικό της ελεγκτή, δεν έχει νόημα να τους κάνουμε να επιλέξουν έναν άλλον, γιατί τον ίδιο θα επιλέξουν τελικά. Αυτό θα αυξήσει απλώς το κόστο και για την επιχείρηση και για τον οικονομικό ελεγκτή και δεν θα προσφέρει τίποτα σε κανέναν. Επίσης, Για μένα αυτό δεν αποτελεί λύση το να γίνει εναλλαγή των επιχειρήσεων. Καλύτερο να κάνουμε εναλλαγή των εταίρων. Θεωρώ ότι ο διτός έλεγχος, ο κοινός έλεγχος, το joint audit, δεν αποτελεί λύση ούτε αυτός θα ήταν δύσκολο να καθιερωθούν ποσοστά. Αυτό λειτουργεί σε κάποια κρατημέλη εξ όσων γνωρίζω, αλλά αποτελεί μόνο μια σύσταση. Ας πούμε ότι έχουμε μια επιχείρηση που έχει φυγατρικές όλα τα κρατημέλη και η σύσταση είναι να επιλέξουν αυτές οι φυγατρικές όποιο οικονομικό ελεγκτή επιθυμούν. Η μητρική εταιρεία δεν επιβάλλει στις φυγατρικές της την επιλογή κάποιου συγκεκριμένου οικονομικού ελεγκτή. Επίσης, κατά την άποψή μου, δεν θα πρέπει να υποχρεώσουμε τους οικονομικούς ελεγκτές να υποβάλουν εκθέσεις στις αρχές. Έχω μελετήσει με τους εμπλεκόμενους παράγοντες και όλοι συμφωνούν ότι αυτό το οποίο επιθυμούν είναι συνεργασία με τους ε, οικονομικούς ελεγκτές, δηλαδή περιοδικές συναντήσεις μεταξύ αρχών και οικονομικών ελεγκτών. Αυτές είναι οι προτάσεις που έχω να υποβάλω μέχρι στιγμής. Θα τις υποβάλω στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Όπως σας είπα, έχω ήδη συζητήσει για όλα αυτά με τους αδέρφους μου στο ΕΛΚ και με άλλους εκτός ΕΛΚ. Θεωρώ Ελπίζω μάλλον ότι κυρίως όσον αφορά την ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να, να αναπτυχθούν, αυτή είναι μια πρόταση που θα την, ε, να την υποστηρίξει η αριστερά και να καταλήξουμε σε έναν επιθυμητό συμβιβασμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία να έχει το λόγο. Ευχαριστώ. φορές ξαφνιάζομαι όταν δεδομένων των εξελίξεων, της παρατήρησης της, ε, των αντιδράσεων των χρηματοπιστωτικών αγορών τα τελευταία δύο χρόνια, ε, εμφανίζεται κάποιος γεμάτος αισιοδοξία στην ε, αρχή και το ιδεώδες της αυτορύθμισης ενός ε, ιδεώδους κόσμου μέσα σε ένα σύνολο λιγοπολίων και εξουσιών και κυριαρχικό κυρίαρχης θέσεως. Δεν μπορώ λοιπόν να ακολουθήσω αυτή την πεποίθηση και δεν νομίζω ότι μπορεί να σα ακολουθήσει και κανεί άλλο, η πλειοψηφία πάντα των μελλον του Κοινοβουλίου. Α μην υπησέλθω σε λεπτομέρειε. Α αναφερθώ πιο συγκεκριμένα σε κάτι το οποίο έχει ε, άμεση σχέση με την έκθεση. Ε, βλέπουμε εδώ μια παρουσίαση μια μελέτη αντικτύπου για τη μελέτη αντικτύπου. Μα, εγώ δεν περίμενα κάτι τέτοιο όμω. Εγώ περίμενα αυτό που προβλέπει και η διοργανική συμφωνία, ότι δηλαδή τα θεσμικά όργανα, μεταξύ άλλων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προβαίνουν σε αξιολόγηση αντικτύπου για τα νομοθετικά κείμενα, αλλά όχι για το η μελέτη αντικτύπου κάποιου άλλου. Μια εν τέλει πολιτική αξιολόγηση για την οποία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σπαταλάμε πόρους. Γιατί αν ήθελα κάτι τέτοιο θα έλεγα, εάν έβλεπα ότι μου λείπει κάτι θα έλεγα να εδώ λείπει αυτό και εκείνο, αλλά δεν μπορώ να ενδιαφέρομαι τόσο πολύ για αυτό που θα πει ένα θεσμικό όργανο στο, δικό μας, ε, το Κοινοβούλιο και στις δικές μας τις υπηρεσίες με ενδιαφέρει σε σχέση με αυτό που επιδιώκει το Κοινοβούλιο, τι ίδιου αντίκτυπο μπορεί να έχει ένα νομοθέτημα. Άρα πρέπει να πω ότι η μεθοδολογία που ακολουθήσατε δεν με ικανοποιεί, δεν αντιστοιχεί σε αυτά τα οποία περίμενα σε σχέση με αυτή τη νέα μονάδα, τη νέα υπηρεσία. Εάν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσουμε, πρόκειται να την αξιοποιήσουμε για να αξιολογήσουμε, να λάβουμε απαντήσεις σε ερωτηματικά που έχουμε εμείς και όχι να λάβουμε κάποιες πολιτικές εκτιμήσεις για τη μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και εμείς τελευταία ανάλυση, θα το κάνει κανείς άλλος για μας. Και στην Επιτροπή Μεταφορών έχω δει ήδη μελέτες αντικτύπου, οι οποίες ε, παρουσίαζαν διάφορους παράγοντες, αυτό θα ήθελα να δω δηλαδή και εν προκειμένου, που μπορεί να επηρεάσουν, ε, που μπορεί να επηρεαστούν από ένα νομοθέτημα. Αυτό είναι το καθοριστικό σημείο. Και γι' αυτό θα πρότεινα να βρείτε ένα διαφορετικό δρόμο, γιατί αυτός που έχετε πάρει είναι λάθος. Ευχαριστώ, κυρία Τάιν. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον συγκεκριτή για το πολύ διεξοδικό έγγραφό του, για το πολύ καλό έγγραφο εργασία. Αποτελεί μια καλή αφετηρία για την αξιολόγηση του εγγράφου της Επιτροπής, αλλά ταυτόχρονα εκθέτει και διαφορετικές ε, ε, αντιλήψεις κατά τρόπο που πιστεύω καλύπτει όλες τις ομάδες, Γιατί θεωρούμε όλοι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος αυτής της Επιτροπής Αξιολόγηση. Το θέμα είναι όμω πώ, σε ποιο βαθμό πρέπει να ενισχυθεί αυτό ο ρόλο και ασφαλώς θα πρέπει αυτή η υπηρεσία αξιολόγηση να μπορεί να επαληθεύει την, ε, τις αξιολογήσεις τρίτων, εκεί δηλαδή όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις από αξιολογήσεις τρίτων που ίσως ήταν μερικές φορές μεροληπτικές και χρησιμοποιούμε μια πιο ουδέτερη θεώρηση. Ο εισηγητής, τουλάχιστον από ό,τι αντελήφθην εγώ, ρητά αναφέρεται προς το παρόν μόνο στα pure audits, δηλαδή τον καθαρό λογιστικό έλεγχο. Αυτό αναφέρει στον γραφό του. Δεν έχω αντίρρηση ως προς την τοποθέτηση αυτή. Αυτή ήταν άλλωστε μέχρι τώρα πάντα η γραμμή των φιλελευθέρων. Αυτό που δεν βλέπω ξεκάθαρα είναι η διαφοροποίηση μεταξύ Ε, μιας επιχείρησης ε, που αφορά ένας έλεγχος, δηλαδή διαφοροποίηση μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αφενός ε, αφετέρου των οργανισμών κοινή ωφελία και κατά τρίτο λόγο μεταξύ αυτών όλων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν έχω αντίρρηση ως προς ε, το γεγονός ότι μια επιχείρηση όπως η Procter Gamble ή η Siemens ε, μπορεί να έχει ε, δημοσιονομική ελεγκτή εδώ και 100 χρόνια και 200 χρόνια δεν με νοιάζει εμένα. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει μια χρηματοοικονομική κρίση δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να ε, υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με μια από αυτέ τι επιχειρήσει. αντίων ε, εάν έχουν καταφέρει να έχουν μια, ένα προσεκτικό έλεγχο και αξιολόγηση και κλειτώσουν την κρίση τόσο το καλύτερο. Εν γέννη για την αξιολόγηση αντικτύπου, όταν επισκεφθήκαμε τι ΗΠΑ, με ενδιαφέρον διαπίστωσα ότι δεν έχουν φτάσει δεν έχουμε φτάσει εμείς μάλλον σε πολύ καλά αποτελέσματα όπως ε, θα θέλαμε τουλάχιστον όπως ήταν η αρχική πρόθεση όταν εισήχθη αυτή η ιδέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να γίνεται αυτή η αξιολόγηση επιπτώσεων ιδιαίτερα στο βέβαια του λογιστικού ελέγχου έχει κεντρική σημασία αλλά σε κάθε τομέα θα πρέπει να γίνεται αυτή η αξιολόγηση επιπτώσεων ε, αντικτύπου και εν γέννη το κοινοβούλιο ή δυνατόν εξωτερικά θα πρέπει, από ανεξάρτητο, δηλαδή, από ανεξάρτητο φορέα θα πρέπει να ε, διεξάγει, να δίνει εντολή για διεξαγωγή μιας ανεξάρτητη ε, μελέτη αντικτύπου. Βέβαια και η Επιτροπή μπορεί να κάνει τη δική τη πλευρά της. πάση περιπτώσει όμω αυτό εξαρτάται και από το σύστημα που θα έχει ο καθένα, γιατί μπορεί να έχει μια Ευρωπα... η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια δική τη μελέτη αντικτύπου που την έχει εδώ και πολύ καιρό ενώ εμεί τώρα μόλι ξεκινήσαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο κακή αυτή η μελέτη αντικτύπου αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία η μελέτη αντικτύπου μπορεί να δώσει διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που δώσει η αντίστοιχη μελέτη αντικτύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλωστε αυτό διευστώνουμε. Και η μελέτη αντικτύπου του Κοινοβουλίου λέει ότι η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σφάλματα, ενέχει σφάλματα. Οι επιλογές δεν αρκούν δεν δίνουν τα απαιτούμενα αποτελέσματα και όπως είπε και ο Μπόντου, διαπιστώνουμε ότι δεν είναι επαρκή η μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν διαπιστώνει σχέση αιτίας και αιτιατού ε, μεταξύ οικονομικής κρίσης και ε, αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Δηλαδή δεν φαίνεται να θεωρεί ότι υπάρχει κάποια ε, ελλειπή συμπεριφορά από πλευρά των δημοσιονομικών ελεγκτών στην ε, ε, όλη κατάσταση και ότι αυτή η ελλειπή συμπεριφορά μπορεί να οδήγησε να επέτεινε την οικονομική κρίση. Αυτά. Τώρα για τις συμβαστικέ τροπολογίες 15 και 16 πρέπει να πω ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία για του δικού μα δημοσιονομικού δημοσιονομικούς γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε μία βάση ώστε αυτοί οι δημοσιονομικοί ελεγκτέ στο μέλλον να μην έχουν μόνο μια περιθωριακή δυνατότητα αξιολόγηση, αλλά να μπορούν να μπουν στην ουσία, δηλαδή να αποφευχθεί αυτό το οποίο η κυρία Λίχτεμπεργκερ έχει επικρίνει στη τελευταία ανάλυση και να έχουν τα συγκεκριμένα στοιχεία από μια μελέτη. Δημοσιονομικό Ινστιτούτο, συγγνώμη, Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο διορθώνω, λέει ο Μιλήτρια, να μην κάνουμε λάθο αυτά που λέμε. Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο, λοιπόν, που στην τελευταία ανάλυση χρειάζεται για να διασωθεί να απορροφήσει χρήματα που διαθέτει ο Ευρωπαίο Προλογούμενο. Αυτό λοιπόν γιατί υπάρχει σαφή σαφής ε, σύνδεσμος μεταξύ του οδηγία ε, για τη, τα λογιστικά πρότυπα, για το δημοσιονομικό έλεγχο, της ε, προκείμενης εδώ συζήτησης και άρα θα πρέπει με τις συμβεστικές τροπολογίες να συζητήσουμε εάν εάν μπορούν να είναι δεκτέ για όλες τις ομάδες. Εγώ σας λέω από τώρα ότι είμαι σύμφωνη. Πρόκειται για ένα βλέμμα στο μέλλον. Φυσικά δεν είναι και το τελευταίο και οριστικό, μπορεί να χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση μελέτη, αξιολόγηση, αλλά αυτό προκύπτει τουλάχιστον από τη μέχρι τώρα φιλολογία. Ε, δεν θα επισέλθω σε περισσότερες διαπιστώσεις προς την αξιολόγηση αντικτύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τι επικρίσει που ακούστηκαν νωρίτερα για την αξιολόγηση αντικτύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα ήθελα εν γέννη να υποστήριξω τη γραμμή που ακολούθησε ο εισηγητή. πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και από πλευρά Γερμανία ε, σημειώνονται διάφορε επεμβάσει στην αγορά. Πρέπει να είμαστε λοιπόν στο δυνατόν πιο προσεκτικοί και διακριτικοί. Είναι ο πιο ασφαλή τρόπο αυτό. Πολλά είναι τα κράτη τα οποία ε, δοκίμασαν τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι λύσει τι οποίε είχε προτείνει, χωρί όμω επιτυχία. Τη δοκίμασαν για ένα διάστημα και μετά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν γιατί ήταν ότι δεν ήταν η σωστή προσέγγιση. Και διαπιστώνουμε θλίψη το αναφέρω μάλιστα διότι το Κοινοβούλιο εδώ και δυόμιση χρόνια ασχολείται με το θέμα αυτό, με τους δημοσιονομικούς ελεγκτές λοιπόν. Ε, η δουλειά λοιπόν του δημοσιονομικού ελεγκτέη σημαίνει σοβαρή δουλειά, σημαίνει πολύ σημαντική υποχρέωση διακριτικότητα, σοβαρότητα, εξαιρετική κατάρτιση και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ακόμη πιο θλιβερό το γεγονό ότι αυτό το σώμα των ελεγκτών, που είναι μικρό σε τελευταία ανάλυση, ευάριθμο, ε, βρίσκεται σε τέτοια κλειδονισμούς και αντιπαραθέσεις εσωτερικές. Και έτσι βρισκόμαστε σε αυτήν την αξιολόγηση αντικτύπου με μια ντάνα ολόκληρη εγγράφων για την αντίστοιχη μελέτη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τα κριτήρια τη Κοπεχάγη και δεν ξέρω με τι άλλο που μα δώσατε. Δηλαδή αυτέ οι έντονες αντιπαραθέσει δεν θα έπρεπε, πιστεύω, να φτάσουν μέχρι εδώ σαν ένα πόλεμο ε, χαρτιού ε, εγγράφων. Ας κοιτάξουμε σε τελευταία ανάλυση πόσο μεγάλες είναι οι προσπάθειες να ε, ε, εξασφαλιστεί η επιρροή στην υπόθεση αυτή ε, Πιέσει ε, Πανταχόφερ θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα πραγματικό πεδίο μαχών. Ε, τα λόμπι είναι παρόντα, η Επιτροπή προσπαθεί να, διατηρήσει την επιρροή τη στην υπόθεση αυτή. Αλλά νομίζω ότι όλε αυτέ οι αντιπαραθέσεις για ένα τόσο βάριθμο, όπω είπα, σώμα δεν αξίζουν πραγματικά, δεν το τιμούν. Είναι πολύ σοβαρό το επάγγελμα που κάνουν και θα πρέπει να είμαστε στο δυνατόν πιο διακριτικοί και να κρατάμε τι αποστάσει μα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, για τα όσα είπατε για τα λόγια πρέπει να πω ότι υπάρχουν ε, πράγματι, είσαστε πολύ ευστοχοί, πολλά στοιχεία. Πολλές επιθέσεις από τα λόμπι. Εν πάση περιπτώσει, πέραν τη ε, αξιολόγηση αντικτύπου, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο ένα καθήκον που έχει αναλάβει η σχετική μονάδα Impact Assessment. Πρέπει να αξιολογεί αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι πολλέ φορέ μέσα στο Κοινοβούλιο εκφράζονται αμφιβολίε για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει αυτή τη μελέτη αντικτύπου. Και έτσι στη Διοργανική Συμφωνία του 2003 λέγεται ξεκάθαρα ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβαίνει σε αυτή τη μελέτη αντικτύπου και εμεί να τη συμπληρώνουμε με τροπολογίες αλλά τουλάχιστον έξι ψηφίσματα έχει διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντωμεταξύ από την περίοδο του 2003 δηλαδή μέχρι τώρα μια πραγματικά ανεξάρτητη μελέτη αντικτύπου, ψηφίσματα τα οποία έχει αγνοήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύο ψηφίσματα τα οποία ζητούσαν τη θέσπιση μια κοινή υπηρεσία σε παραδείγματι. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά γιατί είχαμε ζητήσει και μέσα από τη Διοργανική Συμφωνία να γίνει διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν δέχτηκε ο πρόεδρο τη Επιτροπή, ούτε και τώρα ακόμα το δέχεται. Και έτσι βρέθηκε αυτή η λύση, δηλαδή η δική μα ανεξάρτητη μελέτη αντικτύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που όμω ε, πάλι ε, καταλήγει σε επικρίσεις σοβαρέ για τη μελέτη αντικτύπου από πλευράς Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι κάτι το όχι ασυνηθιστό, πρέπει να σας πω, είναι κάτι το μάλλον το τριμμένο και πρέπει να σας πω ότι και οι πιέσει ε, ει βάρο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενισχύονται, ώστε την προσεχή θητεία να είναι πιο απρόσκοπτη η πορεία προς την ε, λύση για μια κοινή μελέτη αντικτύπου. Εν πάση περιπτώσει θα βρεθεί μια λύση, αλλά τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Λίχτεμπεργκερ ε, και μετά η μονάδα για το impact assessment να μας κάνει την παρουσίασή της. Κυρία Λίχτεμπεργκερ, ναι, θα συμφωνήσω ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα τη μελέτη αντικτύπου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν μέρη, διότι σε ορισμένου τομεί μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολλές οι και ίσως δεν αρκεί να λέμε ότι θα, κάνουμε, θα, θα κοιτάξουμε τι συνέπειες μπορεί να έχει κάτι, πρέπει να κάνουμε μία πρόταση και μετά να δούμε αν αυτή η πρόταση εσπσταθεί και μπορεί να ε, στηριχθεί. Το να γίνει όμως μελέτη αντικτύπου για μία μελέτη αντικτύπου μου φαίνεται μακροπρόθεσμα αντιπαραγωγικό σε να βρισκόμαστε σε ένα μεταεπίπεδο και να αρχίσουμε να χάνουμε σιγά σιγά την επαφή με το στέρεο έδαφος, με τη γη. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρούμε μια πιο ε, προσγειωμένη λύση και θα έλεγα η ανεξαρτησία της μελέτης αντικτύπου θα πρέπει να διασφαλιστεί πολύ σαφέστερα γιατί πια δεν βλέπω να υλοποιείται η απέτηση για την ανεξάρτητη μελέτη αντικτύπου, για την ανεξαρτησία της μελέτης αντικτύπου και επίσης έχω πρόβλημα σε ένα βαθμό μέχρι τώρα ε, ως προς το εξής, ότι τον, να διαβάζω μια έκφραση αντιλήψεων επόψεων για ένα θέμα μου φαίνεται κάπως παράξενο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν είναι έτσι, α μην το λέμε μελέτη αντικτύπου για μια μελέτη αντικτύπου. Α το λέμε γνωμοδότηση επί τη μελέτη αντικτύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει νόημα αυτό που λέτε. Εκεί είναι που δυσκολεύομαι νεολογικά. Γιατί δεν κοιτάμε να κάνουμε μια αντίστοιχη μελέτη αντικτύπου, αλλά κοιτάμε να ελέγξουμε μια μελέτη αντικτύπου κάποιου άλλου που τι είναι, έχει πάει καλά και τι έχει πάει στραβά. Είναι δύσκολο όλο αυτό μου φαίνεται. Τώρα πέραν αυτού τι μπορούμε να κάνουμε. Ίσως να μετατραπεί σε ένα προπέτασμα καπνού το οποίο δεν θα μας επιτρέψει εν τέλει, αν δεν το αντιμετωπίσουμε σωστά όλο αυτό το θέμα, να ε, δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Παρακαλώ για να ακούσουμε και εσάς. Θα προσπαθήσω τώρα να αναλύσω την ανάλυση της ε, μελέτης αντικτύπου. Ε, μετά από αίτημα της Επιτροπής, πράγματι προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα της μελέτης αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα είμαι σύντομη για τα συμπεράσματα, αλλά θα σας εξηγήσω πώς προχωρήσαμε και ποιο ήταν ακριβώς το πεδίο εφαρμογής και ο σκοπός της δουλειάς μας. Γιατί στο έγγραφο, το ενημερωτικό αυτό έγγραφο δεν νομίζω ότι κρίνουμε την ουσία της πρότασης, ούτε τα θετικά στοιχεία των προτάσεων πολιτικής που περιλαμβάνει. Η μόνη ανάλυση την οποία κάνουμε είναι εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην μελέτη αντικτύπου αυτή που είναι ένα γερό έγγραφο 280 σελίδων που συνοδεύει τις δύο προτάσεις, η μελέτη αντικτύπου που συνοδεύει τις δύο προτάσεις έχει χρησιμοποιήσει τις μεθόδους και την ε, λογική που είναι ε, αυτή που χρειάζεται για τη στήριξη των προτάσεων και ελπίζουμε ότι εντοπίσαμε ε, θέματα που αφορούν τη μεθοδολογία και τη λογική τα οποία βοηθούν την Επιτροπή να εντοπίσει τα θέματα που εσείς θέλετε να θέσετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητήσετε περαιτέρω εξηγήσεις ε, για κάποια από τα θέματα αυτά. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι αυτή η μελέτη αντικτύπου σαφώς είναι σημαντική δουλειά. Συνολικά πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα, ε, μια συνεκτική και ουσιαστική αξιολόγηση των περισσότερων ε, προτάσεων. Κυρίως όσον αφορά τις αλλαγές πολιτικής που προτείνει, η τροποποιημένη οδηγία των ελέγχων. Όμως, διαβάζοντας την μελέτη αντικτύπου και συγκρίνοντας ε, συγκρίνοντάς τα, με, την, ε, με τα πρότυπα, τα πολύ ψηλά πρότυπα που έχει θεσπίσει η Επιτροπή για τις μελέτες αντικτύπου, μπορέσαμε να εντοπίσουμε κάποιες αδυναμίες. Ή ότι εντοπίζει σημεία επί των οποίων θα μπορείτε να κάνετε ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν φτάσετε σε όλα τα στοιχεία. Το πρώτο που εντοπίζουμε είναι, που θέλαμε να δούμε μάλλον είναι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπόρεσε ξεκάθαρα και με πιστικό τρόπο να διατυπώσει το πρόβλημα. Το γιατί χρειάζεται παρέμβαση στην αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών, κυρίως δε των επιχειρήσεων του δημοσίου συμφέροντος. Νομίζουμε ότι εντοπίζει τους προβληματικούς τομείς η Κομισιόν που σχετίζονται με τους στόχους της πολιτικής. Άρα εδώ δεν έχουμε πρόβλημα. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι η σειρά των εναλλακτικών πολιτικών που προτείνεται είναι συνεπής με τους στόχους της πρότασης. Αν όμως κοιτάξουμε το κείμενο της Επιτροπής αυτό καθεαυτό είναι σαφές ότι πίσω από αυτούς τους στόχους όπως ας πούμε το να επιτευχθεί το επίπεδο των προσδοκιών να είναι μικρότερο το χάσμα των προσδοκιών από τους ελεγκτές κτλ. Δύο είναι τα κίνητρα της πρότασης. Πρώτον, η έλλειψη, η ε, τα ε, τα, κάποια προβλήματα στην ποιότητα των οικονομικών ελέγχων στην, στην κοινότητα που έχουν ενδεχομένως συνεισφέρει στην οικονομική και τη χρηματοοικονομική κρίση. Αυτό δεν το αμφισβητούμε με, τη, με το εγγραφό μας. Απλώς διερωτόμαστε. Σας έχει δώσει επαρκή στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το στηρίξει αυτό. Το δεύτερο κίνητρο είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στον ανταγωνισμό της αγοράς των οικονομικών ελέγχων. Πιθανώς να υπάρχει, δεν το γνωρίζουμε. Το ερώτημα είναι, με τη μελέτη αντικτύπου της Κομισιόν, το υποδεικνύει την ύπαρξη αυτού του προβλήματος. Και η απάντηση σε αυτά τα δύο ερωτήματα δεν είναι μια θεωρητική άσκηση, διότι μόνο αν το πρόβλημα έχει τεθεί με σαφήνεια. Μπορεί κανείς να αποφασίσει αν οι προτινόμενες λύσεις του θα έχουν θετικό αποτέλεσμα. Αν κανείς είναι ασαφής ε, ως προς το πρόβλημα που θέλει να αντιμετωπίσει, μπορεί να λάβει μέτρα, αλλά αυτά δεν θα στηρίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία, όπως λέει η Επιτροπή ότι θέλει να γίνεται στις νομοθετικές προτάσεις της, που να στηρίζονται δηλαδή αυτές σε στοιχεία. Και βεβαίω το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να έχει τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, για την ε, αιτιολογική σχέση ανάμεσα στις ε, ε, αποκαλούμενες ελλείψεις των, τους ποιότητας του ελέγχου και στην κρίση, Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι δύσκολα μπορεί κανείς να το τεκμηριώσει αυτό απτά. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί πραγματικά να το αποδείξει αυτό. Και απολύτως, είναι απολύτως σαφές σε όλους ότι το η καλή λειτουργία του επαγγέλματος του οικονομικού ελεγκτή θα συνεισφέρει θετικά στην χρηματοοικονομική σταθερότητα. Αυτό είναι διαμφισβήτητο. Τελικά λοιπόν θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι δεν μπορεί να τεκμηριώσει απόλυτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτών των, την ουσιαστική σχέση. Αλλά αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι ότι αυτή η μελέτη αντικτύπου ε, για κάποια από τα μέτρα πολιτικής, τα ε, κάποια από τα μέτρα πολιτικής και μάλιστα από τα πιο αμφιλεγόμενα, τα στηρίζει σε θέματα αγοράς. Βεβαίως οι τέσσερις μεγάλες εταιρείες, έχουν τεράστιο μερίδιο της αγοράς. Αυτό είναι σαφές. Όμως ως δικηγόρος ειδικό στον ανταγωνισμό γνωρίζω ότι τα μερίδια αγοράς από μόνα τους δεν οδηγούν αυτόματα αυτά καθεαυτά σε στρέβλος του ανταγωνισμού. Δεν λέω ότι δεν το κάνουν. Δεν το γνωρίζω. Σε κάποιες περιπτώσεις το κάνουν. Και ίσως σε αυτή την περίπτωση όντως να συμβαίνει αυτό. Αλλά το πρόβλημά μου με αυτή τη μελέτη αντικτύπου είναι ότι δεν μας το αποδεικνύει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το περιγράφει το μεγάλο μερίδιο αγοράς, συγκρίνει με άλλους τομείς και καταλήγει ότι ενδεχομένως υπάρχει πρόβλημα. Αλλά η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού. Έχει τα δεδομένα και τις δεξιότητες ε, για να μπορέσει να αξιολογήσει και να εκτιμήσει την κατάσταση της αγοράς και ε, έχουν ε, εκπονήσει αυτή τη μελέτη αντικτύπου. Και εδώ αυτό το πρόβλημα έχω εντοπίσει, ότι δεν γίνεται δεν αποδεικνύεται αυτό. Αυτό δεν αποτελεί κρίση για το αν και κατά πόσον τα προτινόμενα μέτρα είναι σωστά ή για το αν και κατά πόσον θα πρέπει να το εγκρίνεται αυτό ή εκείνο. Λέμε ότι τώρα, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω διευκρινήσεις από την Επιτροπή σχετικά με την ορθότητα των ισχυρισμών της, ότι δηλαδή αυτά τα μεγάλα μερίδια αγοράς αποτελούν πρόβλημα στον ανταγωνισμό. Και πιστεύω ότι αυτό δεν θα μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να σας το απαντήσει. Μετά τον καθορισμό του προβλήματος είδαμε ε, την αξιολόγηση που αναμένεται από την πρόταση αυτή. Και πάλι για τα περισσότερα μέτρα υπάρχει ξεκάθαρη ανακεφαλαίωση, είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους, καλά τεκμηριωμένα, αλλά για κάποιες προτάσεις, δυστυχώς για τις πιο τα πιο αμφιλεγόμενα στοιχεία των προτάσεων, γνωρίζουμε ποιες είναι η υπεχωρωτική εναλλαγή, οι περιορισμοί της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών, ε, οι, μη... οι αποκλειστικά ελεγκτικές επιχειρήσεις, θεωρούμε ότι η αξιολόγηση αντικτύπου θα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερα κυρίως όσον αφορά το κόστος και τα ωφέλη αυτών των μέτρων που ποτέ σχεδόν δεν ποσοτικοποιούνται. Βεβαίως δεχόμαστε, όπως απαιτείται και από τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές της, η ε, Κομισιόν είναι ανοιχτή και διαφανή ως προς την έλλειψη δεδομένων. Το παραδέχεται ότι δεν μπορεί να σας παράσχει ε, πρόβλεψη για το, πρόγνωση για το κόστος. Όμως, ακόμα κι αν κανείς μπορεί να το δεχτεί αυτό, το αποτέλεσμα είναι ότι γίνεται εξαιρετικά δύσκολο να κρίνει κανείς το πιθανό το πιθανό αντίκτυπο αυτής τη πρότασης γιατί δεν, δίνεται, δεν, δεν δίνονται νούμερα. Να σας δώσω ένα εντυπωσιακό παράδειγμα. Στην απαγόρευση της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στις ε, μονάδες που ελέγχονται, λέει η Κομισιόν, δεν υπάρχει άμεσο κόστο. Ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει. Όμως το έμεσο κόστο υφίσταται, αλλά δεν μπορεί να εκτιμηθεί επειδή εξαρτάται από την γενική αναδιάρθρωση της αγοράς. Αλλά αυτό είναι μια κυκλική <laughs> λογική. Λένε δεν μπορούμε να σας πούμε το κόστος της αναδιάρθρωσης λόγω της αναδιάρθρωσης. Καλά όλα αυτά, αλλά αυτό δεν σας βοηθά, κατ' ουδένα τρόπο δεν σας βοηθά να, καταλήγει, να κατανοήσετε τις συνέπειες της πρότασης. Επίσης θεωρούμε ότι η έλλειψη αυτή μιας ποσοτικοποιημένης ανάλυσης ε, είναι μια έμεση συνέπεια της έλλειψης λεπτομερούς ανάλυσης της αγοράς. Μια άλλη περίπτωση όπου η μελέτη αντικτύπου δεν αντιστοιχεί καν στην πρόταση είναι ο υπολογισμός της περίοδου εναλλαγής. Δηλαδή η μελέτη αντικτύπου αφορά ε, πόσο, θα είναι, πόσο ιδανική θα είναι η εννεαετής περίοδος εναλλαγής. Και ξαφνικά η πρόταση ε, είναι μια πρόταση εναλλαγής εξαετής και μπορεί κανείς να ρωτήσει την Επιτροπή για τη διαφορά αυτή. Από πού, σε τι οφείλεται αυτή η διαφορά. Εν κατακλείδη, εν ένα μέρος τουλάχιστον αυτών των προτάσεων έχουν επικριθεί πολύ από τον κλάδο. Το βασικό πρόβλημα συνίσταται από ό,τι μοιάζει όχι τόσο στους στόχους των προτάσεων, αλλά στην αναλογικότητα κάποιων μέτρων μια ουσιαστική μελέτη αντικτύπου καλύτερα ποσοτικοποιημένη, καλύτερα αιτιολογημένη και με περισσότερα, περισσότερο τεκμηριωμένη θα βοηθούσε να υπερασπιστούμε καλύτερα αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ρωτώ αν υπάρχουν ερωτήσει προς τη μονάδα. Εγώ θα ήθελα για την Επιτροπή κάτι να ρωτήσω. Την πρώτη φορά από την πρόταση αυτή πρώτη μου σκέψη ήταν γιατί την καταθέσαμε την πρόταση αυτή. Εφόσον είναι κάτι το οποίο ρυθμίζεται με την νομοθεσία, αφού υπάρχει μια ισχυρή Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό, υπάρχει γερή νομική βάση για τον ανταγωνισμό, γιατί δεν το ρυθμίζεται με μια νομοθετική παρέμβαση στον τομέα του ανταγωνισμού. Και βεβαίως γιατί δεν γίνεται έρευνα για ενδεχόμενο παράβαση τη σχετική νομοθεσία. Το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει ε, μια διεξοδική μελέτη της αγοράς των συνεπειών κτλ. Και ρωτώ εάν υπάρχει μεσοπρόθεσμα κάποια τέτοια πρόθεση από πλευρά τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Εάν το έκανε αυτό, θα μπορούσε να διαβλέψει κάποιε τάσει των αγορών Γι' αυτό λοιπόν ε, ερωτώ γιατί δεν γίνεται. Υπάρχει κανείς από την Επιτροπή που μπορεί κατά προσέγγιση έστω να μου δώσει μια απάντηση στο ερώτημα αυτό ή μήπως μου απαντήσετε ότι δεν είναι τώρα η στιγμή αλλά αργότερα θα μπορέσετε να μου δώσετε κάποια απάντηση. Κύριε Μπάση. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Λένε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Εμείς μετά τη μελέτη των διαφόρων συνεισφορών προς την πράσινη βίβλο και αφού παρακολουθήσαμε πολύ στενά τη συζήτηση που προέκυψε μετά από την πράσινη βίβλο, είχαμε θεωρήσει ότι το θέμα αυτό πρέπει να το εξετάσουμε από άλλη γωνία και όχι μόνο με τον νόμο περί Και μάλιστα ο στόχος μας δεν είναι στόχοι να καταπολεμήσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε τους επενδυτές και να φροντίσουμε να υπάρχει ανεξαρτησία των ελεγκτών. Μου αρέσει πάρα πολύ η ερώτησή σας, διότι μου επιτρέπει να απαντήσω τουλάχιστον σε μία από τις παρατηρήσεις ε, που έκανε η συνάδελφος που μας παρουσίασε τη μελέτη αντικτύπου. η οποία βασίστηκε στο γεγονός ότι δεν αποδεικνύουμε το πρόβλημα στα πλαίσια του νόμου ανταγωνισμού. Δεν το αποδείξαμε διότι η νομική μας βάση είναι διαφορετική. Είναι μια νομική βάση εσωτερικής αγοράς και δεν μας ενδιέφερε τόσο πολύ το, η οπτική γωνία του ανταγωνισμού. Γι' αυτό ακριβώς και η πρότασή μας είναι βασισμένη σε διατάξεις που δεν αφορούν θέματα θέμη του ανταγωνισμού. Ελπίζω να σας έδωσα ένα πρώτο σχόλιο για τη συνέχεια της συζήτηση. Δεν ξέρω αν θα μου δώσετε και πάλι το λόγο αργότερα ή όχι, διότι αν δεν μου δώσετε το λόγο θα ήθελα επί τη ευκαιρία να πω και ένα-δυο πράγματα για την αξιολόγηση αντικτύπου. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω Ε, για το έργο σας. Παρακολουθούμε πολύ στενά τα όσα έχετε κάνει φυσικά και συμφωνούμε με τα όσα λέτε σε κάποια σημεία βέβαια, διαφωνούμε με κάποια άλλα. Αυτό όμως το οποίο έχει σημασία και πρέπει να επισημάνουμε ευθύ εξ αρχή είναι ότι ε, ελπίζουμε να συνεργαστούμε με το συνήθι τρόπο με τους δύο συνομοθέτες ώστε να καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για όλους. Αυτό αποτελεί το εφαλτήριό μας και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να το επενθυμίζουμε πάντα. Μας ικανοποιεί επίσης ιδιαίτερα και αυτή η νέα εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για τη Γενική Διεύθυνση Αξιολογήσεων Αντικτύπου, διότι εμείς δεν θεωρούμε ότι τις έχουμε μονοπόλιο της αξιολογήσεις αντικτύπου, δεν θεωρούμε ότι είναι τέλειο το έργο μας, δεν θεωρούμε ότι είναι τέλειο το έργο μας όταν κάνουμε μια πρόταση, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε πάντα διατεθειμένοι να το βελτιώσουμε με τη βοήθειά σας. Δεν θεωρούμε ότι ε, κάνουμε τέλειο έργο όταν κάνουμε μια μελέτη αντικτύπου. Ε, είμαι βέβαιος λοιπόν ότι με τη βοήθεια των άλλων ε, θεσμικών οργάνων, σήμερα το Κοινοβούλιο, αύριο μακάρι και με τη βοήθεια του Συμβουλίου, αλλά Ελπίζω ότι στο τέλος θα καταφέρουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ε, ε μας ε, χαροποιούν οι επικρίσεις σας, μας χαροποιεί το γεγονός ότι γίνεται δουλειά που αφορά το δικό μας το έγγραφο και προσβλέπουμε και στη δική σας την αξιολόγηση για την πρόταση, εάν θέλετε να κάνετε αξιολόγηση, ή προ τι τροπολογίε που θα προτείνετε. Διότι η μελέτη αντικτύπου, κατά την άποψή μου, δεν είναι αυτό σκοπό. Απλώ ε, στόχο έχουν να συνεισφέρουν στην καλύτερη χάραξη πολιτικής και στην καλύτερη νομοθεσία που μπορούμε να ετοιμάσουμε όλοι μαζί. Δεν ε, θα απαντήσω ε, αναλυτικά σε όλες τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που ετέθησαν, όχι γιατί θεωρούμε ότι έχουμε κάνει εμείς την τέλεια δουλειά, αλλά γιατί είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και ε, στο διάλογο για τη μελέτη αντικτύπου και περιμένουμε να γίνει διάλογος μόνο γι' αυτό, επί τη βάση της δικής σας αξιολόγησης. Επιτέλους κάποιος μας βοηθάει και μας γι' αυτό το τόσο δύσκολο καθήκον. Θα το δείτε αυτό όταν θα αρχίσετε να κάνετε πραγματικές μελέτες αντικτύπου και δεν θα επικρίνετε απλώς τις ε, μελέτες των άλλων. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα καταλάβαμε, τα και σας υποστηρίζουμε στα όσα μας είπατε. Δεν βλέπω να στείλει κανείς άλλο το λόγο στο θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης. Να στο κλείσουμε. εκτός και αν θέλει ο κύριο Καρύμ να πει κάτι ακόμα. Παρακαλώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι απίλαυσα την συζήτηση. Ήταν έντονες οι αντιπαραθέσει απόψε. Βρετανική ονείροξη θα το έλεγα. Κύριε Μάσομ, εσείς είσαστε σε μια ζεστή χώρα, ξηρή χώρα και έτσι δεν γνωρίζετε τι σημαίνει wet dream στα αγγλικά, δηλαδή ονείροξη, που είναι πολύ γνωστό σε εμάς με το προχειρό μας κλίμα. Δηλαδή, θέλετε, να αναζητήσουμε τα στοιχεία, τα αποδεικτικά, τα οποία αιτιολογούν μια πολιτική επιλογή. Μα ακριβώς αυτό είναι που, ε, επικρίνουμε, είναι ότι δεν υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία εγκαίρως, δηλαδή ότι γίνεται δουλειά αντίστροφα από ό,τι θα έπρεπε να γίνεται πραγματικά. Και με τα δεδομένα και τα στοιχεία τα οποία μου προσφέρει αυτό το έγγραφο και πρέπει να υπενθυμίσω ότι είναι η πρώτη φορά που αξιοποιείται από εμά αυτή η διαδικασία και πρέπει να πω ότι με προσέφερε αρκετή ικανοποίηση αυτή η δυνατότητα διότι, διότι εγώ ήμουν εκείνο στην Επιτροπή μας, πρέπει να σα υπενθυμίσω, ο οποίο ηγήθηκε της ε, πίεσης για μια διαφανή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και όχι και κλεισμένο των θυρών. Τα σχόλια τα έκανα, τις προτάσεις, χωρίς να έχω καμιά ιδέα για το πού θα μας οδηγήσουν τα πορίσματα αυτής της έκθεσης. Άρα, νομίζω ότι είναι λίγο άδικο να αντιστρέφουμε τους όρους τώρα. Ε, μα πρόεδρος, όχι, όχι, όχι, δεν θα τα πω. Δεν θα σας ε, παρουσιάσω έναν από τα σημεία από τα όσα είπαν οι συνάδελφοι για τον κύριο Μπόντου, για την κυρία Τάινερ. Όντω ε, όντως είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι προτάσεις τους. Περιμένω πότε θα μας δοθεί ευκαιρία να κάτσουμε μαζί να τα συζητήσουμε. Όταν θα έχετε πολύ απτές ιδέες να τις συζητήσουμε και να κοιτάξουμε γραμμή-γραμμή πώς θα συντάξουμε το κείμενο, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ε, πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε κάποιες από τις ιδέες τις οποίες έχετε διατυπώσει, έχετε υπόψη. Η κυρία Λιχτινμπέργκερ έκανε κάποια γενικά σχόλια για την αξιολόγηση αντικτύπου δεν θέλω να επαναλαμβάνουμε πρόεδρε, αλλά είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνουμε αυτό το έργο, αυτή την ε, προσπάθεια. Και δεν θέλω να πω ότι με ευγνώμων προς την ε, υπηρεσία αξιολόγηση αντικτύπου για όλη τη δουλειά και βέβαια για την παρουσία του σήμερα εδώ. Μας δίνουν τις, εξελί, τις εξηγήσεις, τις όπως το έπραξαν. Ε, και πρέπει βεβαίως τη διαδικασία αυτή να την αντιληφθούμε ως μια διαδικασία σε εξέλιξη. Θα ήταν λάθος να θεωρούμε ότι είναι παγιωμένη Πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα προχωρήσει, πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιδέα που είχαμε. Πολύ σύντομα, παρατήρηση της Επιτροπής. Πρέπει, πιστεύω, να γνωρίσουν οι συνάδελφοι ότι είχα καλέσει τον Επιτροπό Μπον και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί δύο φορές μάλιστα προτάσεις έτσι ώστε και εμείς και η Επιτροπή, ίσως και το Συμβούλιο δυνατόν, να καταλήξουμε σε ένα σύνολο προτάσεων που να εξασφαλίζει στο δυνατόν καλή και εδρεωμένη συμφωνία. Ε, διαφορετικά χάνουμε χρόνο. Είχα λοιπόν αυτές τις ε, συζητήσεις, τις επικοδομητικές, ώστε να υπάρξει άλλη μια ευκαιρία για συνάντηση και πρέπει να πω ότι Ξέρω ότι δεν πρόκειται να ικανοποιήσω τους πάντες όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, αλλά δεν επιδιώκω κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλω είναι να έχω ένα καλό σύνολο προτάσεων, μια γερή βάση για να κάνουμε στο δυνατόν καλύτερη δουλειά, βασικά για τους ψηφοφόρους μας. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα μπορούμε να αφήσουμε το σημείο αυτό για να προχωρήσουμε στα συζήτηση των 32 και 33. Νομίζω μπορούμε να τα δούμε ως ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η κυρία Μακάρτη είναι η πρώτη στη σειρά με το υπαριθμό 32 θέμα στην ημερήσια διάταξη και θα συνεχίσω εγώ με το δικό μου. Κυρία Μακάρτη, θέλεις να ξεκινήσετε εσείς. Θα ήθελα να είμαι σαφής, κύριε Πρόεδρε. Θα παρουσιάσω την εκθεσή μου, αλλά μετά θα περιμένω και να μιλήσω ως σκιώδης ο ε, των σοσιαλιστών για τη δική σας έκθεση. Εντάξει, ας το κάνουμε έτσι. Θα κάνω το δικό σας, μετά θα ακούσω τι θα πούν οι άλλοι και μετά θα κάνετε εσείς και θα επανέλθω ως εκπρόσωπος των σοσιαλιστών. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που ξοδέψατε για να υποβάλλετε τροπολογίες. Όπως ξέρετε, είχαμε αποφασίσει να μην γίνει ψηφοφορία μέχρι τη σύνοδο του Σεπτεμβρίου και άρα έχουμε χρόνο να σκεφτούμε τα θέματα αυτά. Έχω όμως κάνει κάποιες ε, συμβιβαστικές προτάσεις που θεωρώ ότι αντικατοπτρίζουν την πλειοψηφία των θέσεων που διατυπώθηκαν στην Επιτροπή. Τα γενικά θέματα ασχολήθηκαν με το θέμα της ε, των εκθέσεων αναχώρα ε, επίσης για τις, ε, τα θέματα που αφορούν τις εξορυκτικές, ε, τον εξορυκτικό κλάδο και επίσης ε, οι τροπολογίες της Επιτροπής Οίκων ήταν πιο χαμηλά από ό,τι στην αρχική πρόταση της Κομισιόν. Και λέω ότι δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτά τα ε, χρηματοοικονομικά όρια, αλλά τελικά θα καταλήξουμε με κάποια από αυτά. Κάποια θα έχουμε. Άρα χρειάζεται μια διαπραγμάτευση στο πλαίσιο των ε, τροπολογιών που έχουν ε, υποβληθεί στην δική μου έκθεση και στην έκθεση του κυρίου Λέινε. Όμως σημασία έχει το πιο σημαντικό να συμφωνήσουμε για το τι θα αναφέρουν οι εκθέσεις. Δηλαδή θα είναι εκθέσει σε επίπεδο έργου, σε επίπεδο κυβέρνησης, όπως ε, αναφέρει το, η πρόταση του Συμβουλίου. Και νομίζω τα περισσότερα μέλη δεν συμφώνησαν επ' αυτού. Γι' αυτό οι συμβιβασμοί μου πάνε προς την κατεύθυνση του Συμβουλίου. Υπάρχει όμως πιστεύω περιθώριο για βελτίωση στο τομέα αυτό και επίσης περιθώριο για περαιτέρω συμβιβασμό. Ε, επειδή η πλειοψηφία των ανθρωπολογιών ε, ε, έμοιαζε να συμφωνεί ότι χρειάζεται ένα ε, ετήσιος ισολογισμός της ε, εκθέσεις χώρα και πάλι όμως οι συμβιβασμοί αναφέρονται στις, στη φορολόγηση και στις αποκάλυψη των πληροφοριών. Όταν θα έρθουμε στη δική σας έκθεση, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι θα δούμε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και να βρεθεί συμφωνία. Μετά θέλησα να μελετήσω το θέμα της ε, ελάχιστης ή της μέγιστης εναρμόνισης για τις απαιτήσεις της υποβολής εκθέσεων Ε, κάποιοι ήταν ε, πολύ κατά της ε, μέγιστης εναρμόνισης, άλλοι ήταν πολύ κατά της ελάχιστης. Τα κράτη-μέλη μπορούν, σύμφωνα με τις προτάσεις μας, να επιβάλλουν επιπλέον οι προϋποθέσεις τη μικρομεσαία Γιατί και στις δύο εκθέσει έχουμε συμφωνήσει ότι θέλουμε να περικόψουμε τη γραφειοκρατία. Αλλά βεβαίω είναι έκθεση διαφάνειας, οπότε πρέπει να έχουμε ένα αποδεκτό επίπεδο διαφάνειας και ε, υποβολής εκθέσεων για τις ε, επιχειρήσεις. Και η εμπειρία μου με τις μικρέ επιχειρήσει είναι ότι του αρέσουν οι ρυθμίσει, θέλουν να υπάρχουν ρυθμίσει, αλλά δεν θέλουν να έχουν πλήρη εξαίρεση, γιατί θεωρούν ότι αυτό είναι σημαντικό για τη δική του αξιοπιστία. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα μπορούν να επιβάλλουν περισσότερε, αυστηρότερε απαιτήσει υποβολή εκθέσεων σε μεγαλύτερε επιχειρήσει κατά, κατά την άποψή του. Επίσης, έγινε μια συζήτηση στο Συμβούλιο που αφορά τις ε, εξαγορές και μοιάζει ότι και εδώ μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό. Ξέρω ότι υπήρξαν ανησυχίε για την ε, ε, ανάθεση στην ΕΣΜΑ έγινε μια συζήτηση και προσπάθησα τις ανησυχίες αυτές να τις λάβω υπόψη μου και ελπίζω ότι θα μπορέσει να υπάρξει ένα συμβιβασμό στο σημείο αυτό ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κατευθυντήριες γραμμές ε, Προ αυτήν την κατεύθυνση σε σχέση με το να θεσπίσουμε αυστηρούς κανόνες. Κάποια κράτη-μέλη θέλουν να μπορούν να εκδώσουν κάποιε συμπληρωματικέ κατευθυντήριε γραμμέ. Λοιπόν, ε, αν αυτό γίνεται, τότε τα κράτη-μέλη μπορεί να το κάνουν υποβορφή συμπληρωματικών κατευθυντηρίων γραμμών, αλλά πρέπει να φροντίσουμε αυτές να είναι να έχουν μια αναλογικότητα και να λαμβάνουν υπόψη τους το βάρος που επιβάλλει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, το ε, θέμα της αναφοράς XPRL. Εξ όσων αντιλήφθηκα, αυτό ήταν σημαντικό. Όμως όπως έκανε και ο πρόεδρος με τους κανόνες λογιστικής, θεωρώ ότι εδώ θέλουμε να έχουμε μια ενιαία ηλεκτρονική μορφή υποβολής εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτή τη στιγμή θα, πρέπει να πούμε ότι θα εισάγουμε αυτή την ενιαία ηλεκτρονική μορφή και από εκεί και πέρα θα λάβουμε και πάλι ε, υπόψη μας αν θα μελετήσουμε αν αυτή η μορφή XPRL είναι η κατάλληλη. Αν ναι, θα το κάνουμε και θα το επιβάλλουμε. Αλλά δεν το έκανα από αυτή τη στιγμή, γιατί όπως είπα στους συναδέλφους, γίνονται κάποιες έρευνες αυτή τη στιγμή που λένε ότι υπάρχει υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να αλλάξουν το XPRL, ε, δηλαδή θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν ηλεκτρονικές εκθέσεις, αλλά θα αλλάξουν κάποια στοιχεία. Δηλαδή να μην επιβάλλουμε κάτι το οποίο μετά θα, το, θα ξεπεραστεί από την τεχνολογία και μόνο. Θα ήθελα να δω μια μελέτη αντικτύπου για τις διαφορετικές μορφές υποβολής εκθέσεων όπως τους έχει δοκιμάσει η SCC και μου είπαν διάφοροι συνάδελφοι ότι δεν έχει, δεν έχει γίνει υποχρεωτική η XPRL στην, ε, στις ΗΠΑ παρά μόνο μετά από κάποιο διάστημα χρήσης και δοκιμών. Ε, ένας άλλος συμβιβασμός ήταν το προσαρμοσ... ο... Η... ο προσαρμογή του υπολογισμού των δικαιωμάτων ψήφου είναι σωστό να ενσωματωθεί με τον τρόπο που το κάνω στο συμβιβασμό. Συμφωνεί και με την νομοθεσία που έχουμε ήδη ψηφίσει για το short selling. Άρα το θεωρώ συμπληρωματικό με αυτό. Τώρα, όσον αφορά τις κυρώσεις, και πάλι αυτό είναι ένας τομέας στον οποίο συζητήσαμε. Είδα τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν και όπως σας είπα πριν, ποτέ δεν είμαι ιδιαίτερος ευτυχής όταν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες οικονομικές κυρώσεις γιατί η κατάσταση είναι διαφορετική στα κράτη-μέλη. Αυτό που είναι σωστό στην Βουλγαρία και τη Ρουμανία δεν είναι κατά ανάγκη σωστό ε, στη Γαλλία. Πρέπει να φαίνεται αυτό. Κάναμε καλή συζήτηση με την ε, Επιτροπή και τους συναδέλφους και θα κρατήσω την αναλογικότητα εδώ με κάποιες επιπλέον διατάξεις για τα ε, δικαιώματα ψήφου. Αυτά θα ανασταλούν μετά από, αφού ξεπεραστεί ένα όριο και σε πιο ακραίες περιπτώσεις. Υπάρχει μια λογική εδώ. Επίσης θεώρησα ότι είναι σωστό να πούμε ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον μέτρα και κυρώσεις στα ανώτερα επίπεδα από ό,τι προβλέπει η οδηγία. Και αυτό ε, ακριβώς αντικατοπτρίζει τα διαφορετικά συστήματα θα υπάρξει δηλαδή κάποια ευελιξία και σε αυτούς τους τομείς. Θεωρώ ότι τα επίπεδα που προτείνει η Κομισιόν, τα μέγιστα ή τα ελάχιστα επίπεδα κυρώσεων που πρέπει να επιβληθούν, είναι σωστό να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη που έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα να τα ανεβάσουν. Έχει αυτό μια λογική και αποφάσισα να το υποστηρίξω αν δείτε το, τις συμβαστικές τροπολογίες θα δείτε ότι έχω, κάνει κάποιες, έχω μετακινήσει κάποια. Για την δημοσίευση των κυρώσεων. Θεωρώ ότι αυτή η δημοσίευση των κυρώσεων είναι σημαντική για την αποτροπή των, κρατών μελών να μην δηλαδή να, να μην συμμορφωθούν. Βεβαίως θα περιορίσουμε τις περιπτώσεις όπου δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται οι κυρώσεις, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε ο καθένας που μπορεί να βρει ένα καλό ε, δικηγόρο να μπορεί να το αποφύγει. Είναι σημαντικό να μπορούμε να ενημερώνουμε την κοινή γνώμη και τα μέσα των μέσων ενημέρωσης για αυτούς που δεν ε, λειτουργούν σωστά, γιατί αυτό αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα και αυτό είναι και ένα άλλο ταμέα στον οποίο εργάζομαι, γι' αυτό μπαίνω βγαίνω στην αίθουσα, είναι ο κανονισμό για την κατάχρηση αγορά. Όταν μπορεί κανεί να δημοσιεύσει τα πρόστιμα και τι ποινέ που έχουν επιβληθεί, τότε ε, οι άνθρωποι αρχίζουν να διαρωτώνται τι θα τους συμβεί, θα διαπομπευθούμε, δεν μας αρέσει η διαπόμπευση κλπ. κλπ. Άρα είναι ένα καλό θέμα, αλλά και εδώ έχω κινηθεί προς την κατεύθυνση, λίγο προς την κατεύθυνση της Επιτροπής. Τώρα, η ρήτρα επανεξέτασης. Έχω λάβει υπόψη μου τις προτάσεις της Επιτροπής Οίκων και Διεθνούς Εμπορίου στο κείμενο αυτό και πάλι ζήτησα δύο χρόνια μετά την εφαρμογή της, να την επανεξετάσουμε. Υπάρχει βεβαίως και η δική σου σας ε, έκθεση, κύριε Πρόεδρε, που θέτει κάποια όρια. Όλοι αυτοί είναι τομεί που πρέπει να επανεξεταστούν και πιστεύω ότι η διετία είναι επαρκές διάστημα για να γίνει μια πρώτη έκθεση στο χώρο αυτό. Ας, πρέπει να δούμε και θέματα της εξαίρεσης κάποιων τα υπάρχουν τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι Εθνικές Τράπεζες των κρατών μελών. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες εξαιρέσεις, αλλά μόνο εάν υπάρχει μια έκθεση που να μας ενημερώνει για τον αντίκτυπο αυτών των εξαιρέσεων. Ε, γίνονται λοιπόν, θα υπάρξουν αναθεωρήσεις ε, καθώς συντάσσονται τα ε, θεσμικά πρότυπα. Υπάρχει αυτό η πρόταση της Επιτροπής Οίκων και η εφαρμογή των κυρώσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί τη διετία. Λοιπόν, ζητώ από του συναδέλφου, επειδή ξέρω δεν έχουν το χρόνο το να μελετήσουν τι συμβιβαστικέ τροπολογίε που υπέβαλα, καθώς θα συζητούμε την έκθεσή σας για τα λογιστικά πρότυπα, αυτά είναι ε, σημαντικά για μένα υπάρχουν και άλλοι ε, συμβιβασμοί και κείμενα επ' αυτού. Οι, δικές, οι δικοί μου συμβιβασμοί πόρο απέχουν από τους συμβιβασμούς στο δικό σας κείμενο. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα ευθυγραμμίσουμε τα κείμενα ή τελικά θα πρέπει να ψηφίσουμε. Νομίζω όμως ακούσουμε, ας ακούσουμε τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι από αυτόν και μετά θα πάρω το λόγο ως ομάδα S&D ε, επ' αυτού. Ευχαριστώ. Ωραία, χαίρομαι που αναφερθήκατε στη διαδικασία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε, έχουμε λίγο χρόνο να ασχοληθούμε με τις συμβαστικές τροπολογίες. Σεπτέμβριο το πολύ πολύ μέχρι τα τέλη στο Στρασβούργο μπορούμε να έχουμε κάποια ευκαιρία να συζητήσουμε αν υπάρχει περιθώριο για συμβαστικές τροπολογίες, αν τα καταφέρουμε, αν όχι, επιφασίσουμε το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε να, να συνεχίζεται αυτή η ασάφεια. Πρέπει να τα κλείσουμε τα θέματα αυτά στο βαθμό που μπορούμε. Τώρα, αν μου επιτρέπετε να πω και εγώ δύο λόγια για την οδηγία περί διαφάνειας, διότι απευθύνεται, έχει πολύ μεγάλη σημασία απευθύνεται σε ένα πολύ μεγάλο κύκλο επιχειρήσεων Βέβαια, σε στενότερο ίσω ε, κύκλο από ότι η οδηγία για την ε, υποχρέωση λογοδοσία και τα λογιστικά, το accounting, τη λογιστική, ε, ίσως είναι μία σειρά θεμάτων της οδηγίας της διαφάνειας για μένα ως σκιώδη συγκητή εκ μέρους της ομάδας μου πολύ πιο ευχαίρες να τα χειριστώ όλα αυτά τα θέματα από ότι ως κύριος ως αρμόδιος για την άλλη οδηγία για το accounting. Για το ΕΣΜΑ λοιπόν έχω μια κάπως πιο στενή αντίληψη της κατάστασης, κάπως πιο συσταλτική για τις εκθέσεις καταστάσεως. Αν μπορούν τα κράτη-μέλη να επεξεργαστούν επιπλέον κριτήρια, υπάρχει το ενδεχομένο ο κίνδυνος να επικρατήσει περαιτέρω σύγχυση. Επομένω, θα πρέπει να βρούμε μια πιο προσεκτική τοποθέτηση για το XPRL ως έγγραφο συμφωνώ μαζί σας έχει νόημα ένα τέτοιο σύστημα αλλά πρέπει να δοκιμαστεί πρώτα και να δούμε εάν είναι το καταλληλότερο όντως πάντως ένα τέτοιο ε, electronic reporting format δεν ε, με ενοχλεί εμένα. Νομίζω ότι είναι κάτι το καλό και το βλέπουμε και στα δύο κείμενα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Στο ζήτημα της, ε, των κυρώσεων και την αποζημίωση περίπτωση ποινική ευθύνη. Χαίρομαι για τη διαγραφή των προτάσεων. Ε, για τον τομέα country by country, η συμβαστικές τροπολογίες που προβλέπονται εδώ. ακολουθούν κάποια κριτήρια. Αυτό μπορεί να έχει κάποιες, ε, κάποια πλεονεκτήματα ή και μειονεκτήματα. Πρέπει να το κρίνουν ασφαλώς οι συγητέ, ε, σκιώδης και μη. Υπάρχουν κάποιες προποθέσει που απαιτούνται για κάθε ε, έναν που δημοσιεύει λογαριασμούς. Ίσως θα πρέπει να δούμε αν αυτά θα ισχύουν για όλους τους PIEs ή αλλιώς θα δώσουμε μια διαφορετική λύση. Για το project by project και ιδιαίτερα, ιδιαίτερα στην εξόριξη ε, πόρων από το υπέδαφος είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δει η Επιτροπή, μη γραφειοκριτικά βέβαια πρέπει να ρυθμιστεί το σύστημα για να είναι και αποτελεσματικό για τις ε, εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις. Νομίζω ότι οι προτάσεις είναι καλές, αν και μπορούμε να δούμε μια διαφορετική προσέγγιση σαν δυνατότητα από αυτή που προβλέπει οδηγία για την τήρηση λογιστικών βιβλίων, για το accounting δηλαδή. Αυτά επί το πλήστον και θα ήθελα να συμπληρώσω κάποια στοιχεία σε σχέση με τις δικές μου συμβαστικές τροπολογίες για το accounting, για τα λογιστικά βιβλία, βλέπω ότι σε πολλά από τα θέματα που έχουμε συζητήσει έχουμε προσανατολιστεί αντίστοιχα με αυτά τα οποία συζητεί το, κοινοβου... το Συμβούλιο και στο οποίο υπάρχει δυνατότητα για συμβιβασμούς από ό,τι φαίνεται, αποδεκτούς και για μας. Όχι σε όλους τους τομείς, αλλά σε κάποιους από αυτούς τους τομείς μπορούμε νομίζω να βρούμε λύσεις Εμπνεόμενη, θα έλεγα από αυτά τα οποία έχει συζητήσει και το Συμβούλιο. Η πρώτη συμβαστική τροπολογία έχει να κάνει με μια αιτιολογική σκέψη που μπορεί να αποτελέσει βοήθεια για ερμηνεία. Στην συμβαστική τροπολογία 2 υπάρχει η ιδέα στο corporate governance και corporate social responsibility, δηλαδή ε, διοίκηση επιχειρήσεων και κοινωνική ευθύνη επιχειρήσεων, πρέπει να γίνουν προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην τρίτη συμβαστική τροπολογία είναι το XPRL, αντίστοιχη γραμμή με αυτή της κυρίας Μακάρτη. Στη συμβαστική τέσσερα έχουμε το small regime, δηλαδή προτάσεις αντίστοιχες με αυτές των Γάλλων συναδέλφων, αλλά και άλλων, που είχαν καταθέσει τροπολογίε, δηλαδή μια ευελιξία κατά 20% πάνω κάτω. Αποδεκτό όριο για μένα, αποδεκτή συμβαστική τροπολογία, ώστε να έχουν περιθώριο ελιγμών ε, τα κράτη-μέλη, χωρίς όμως και να χάνεται τελείω η δυνατότητα τη εναρμόνιση. Η συμβαστική 5 αφορά τεχνικού χαρακτήρα προσαρμογές, ε, είναι της κυρίας Κάστεξ ε, λίγο πολύ οι προτάσεις, η συμβαστική έξι, εναλλακτική αξιολόγηση χρηματοπιστωτικών μέσων που επιτρέπεται με βάση και τις ε, οικονομικές συνθήκες να αξιοποιηθούν, αλλά σημειώνω ότι θέλω στο δυνατόν λιγότερα δάνεια του EFS να περιληφθούν μέσα στην έκθεσή μου. Συνειδητά το κάνω αυτό. Συμβαστική 8 αναφορά στην ε, συμβαστική λύση του Συμβουλίου αλλά και μια προσπάθεια εναλλακτική ε, για τη διατύπωση των ισολογισμών ε, στην 9 και τη 10 μετά. Το goodwill, κάτι το οποίο έχει εξετάσει και το Συμβούλιο και που μπορεί να γίνει αυτό και από το Κοινοβούλιο. Στην 11 έχουμε μόνο μία προσαρμογή των ε, διατυπώσεων της 7 και 8 στη 12 μόνο αριθμός εργαζομένων και στη 13 προθεσμία μη δεσμευτική ε, για τα κράτη-μέλη, γιατί σε τελευταία ανάλυση νομίζω ότι είναι διοικητικό μέτρο. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν την ελευθερία να κρίνουν, δεν πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να θεσπιστούν δεσμευτικά όρια. Στην 14 συμβαστική τροπολογία έχουμε την εξαίρεση τη υποχρέωση λογιστικού ελέγχου για τι μικρότερε επιχειρήσει ένα θέμα το οποίο πρέπει να σε απασχολήσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι, γιατί το έχουμε ξανασυστήσει αυτό και με τις ε, μικροεπιχειρήσεις, ε, ε, δεν είναι κάθε μεσαία επιχείρηση επιχείρηση που χρειάζεται διαφορετική μεταχείριση. να σταει μια πίστοση και η τράπεζα την υποχρεώνει να κάνει αυτό και εκείνο, έναν εσωλισμό, έναν λογιστικό έλεγχο, τότε τον προχωρεί και τον υλοποιεί. Ε, ίσως λοιπόν δεν χρειάζεται πάντοτε να έχουμε αυτή την εξαίρεση. Αυτός είναι ο λόγος συμβαστικής πρότασης. 15 Πάλι πάει στην πρόταση του Συμβουλίου και την ε, οδηγία για τον ε, λογιστικό έλεγχο. Το country by country reporting στη συνέχεια. Πάλι παρακολουθώ τα κράτη-μέλη. Δεν είχε προταθεί αρχικά μια έκθεση, μια, ένα σχέδιο εκθέσεως, το εισάγουμε εδώ με την συμβαστική τροπολογία στη συνέχεια και εδώ έχω μια διατύπωση καλύτερη από το αρχικό κείμενο πιστεύω γιατί μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες συμβάσεις για δε τις ποινικέ διατάξεις εισάγω μία ρήτρα grandfather δηλαδή μια ε, ρήτρα μία αναδρομικότητας ώστε να αντιμετωπιστούν ε, ενδεχομένες εξελίξεις στην ε, νομοθεσία αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί και θα απασχολήσει και στο μέλλον τους σκιώδης συγκητές συζητήσεις τους. Payments στη συνέχεια, pipeline transit fees, υπηρεσίες ασφαλείας, πρόσβαση στις πληροφορίες, στα δεδομένα, αριθμός των εργαζομένων, πρόστιμα για ε, περιβαλλοντική ρήπανση, παραδείγματα και άλλα αντίστοιχα συμβαστική λύση για την πρόταση της ενοποίησης στο country by country όταν έχουμε θηγατρική που ενεργοποιείται σε δραστηριοποιείται σε διαφορετικά κράτη-μέλη και μια ρήτρα αναθεώρησης review clause που πάλι έχει ε, ευρεία διατύπωση. Δεν προτείνω, αν και ξέρω ότι ίσως κάποιοι συναδελφοί θεωρούν ότι πρέπει να συμβεί κάπως διαφορετικά, ε, διεύρυνση επέκτηση σε διάλους τομείς, θα δούμε με τους και αν υπάρχει δυνατότητα και δεν έχω προβλέψει επαλήθευση αυτής της ε, έκθεσης, audit, Πράγμα το οποίο ίσως στην περίπτωση της οδηγίας για τη διαφάνεια να ισχύει διαφορετικά, αλλά εδώ, εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ε, η ε, οδηγία για το accounting και όχι επιλεκτικά όπως αυτή για, το, για τη διαφάνεια. Πρέπει να ισχύει για μικρές και μεγάλες, δεν μπορούμε να πούμε ότι εξαιρούνται κάποιες και να ισχύει μόνο για τις πολύ μεγάλες. Αυτό σημαίνει ότι και οι εταιρείε τις οποίες πρέπει να ελέγξουμε σοβαρά θα ελεγχθούν, αλλά και με την ε, ιδέα του παρεπίπτωτος ελέγχου κάποιες που δεν είχαμε υπόψη μας να ελέγξουμε, μπορεί να βρεθούν, να πιάσουν στα δίχτυα. Ε, θα δούμε με την κυρία Μακάρτη πώς θα προχωρήσει η κατάσταση μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Θα βρούμε, πιστεύω, σημεία επικοινωνίας και συμβασμού. Εάν όχι, εάν όχι τότε θα ξανασυστήσουμε το θέμα αυτό και θα ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο στην Επιτροπή μας. Και θα δούμε μετά τι θα βγει μέχρι την Ολομέλεια, η οποία θα κρίνει το βασικό ζήτημα της εντολής του Κοινοβουλίου, το εάν θέλουμε να το χειριστούμε το θέμα αυτό με διαπραγμάτευση, αν θα πρέπει να κλείσουμε την πρώτη ανάγνωση και να περιμένουμε τη δεύτερη με τις θέσεις του Συμβουλίου στην πιο τυπική διαδικασία. Αυτά είχα να σας πω. Η κυρία Τάιν έχει στο λόγο, μετά η κυρία Μακάρτσι, μετά ο κύριο Χέφνερ. Παρακαλώ. Κυρία Τάιν. Εάν σα καταλαβαίνω καλά, κύριε Πρόεδρε, για τι συμβαστικέ τροπολογίε, συζητάμε τώρα, έτσι, τη κυρίας Μακάρτη πρώτα, μετά για σα. Ωραία. Λοιπόν, για την ε, γνωμοδότηση για τις προτάσεις ε, συμβαστικών τροπολογιών για την οδηγία για τη διαφάνεια. Πολύ πρόσφατα τις έλαβα μόλις εχθές και έτσι δεν μπορώ παρά ε, γενικόλογα να τοποθετηθώ. Με την υπαριθμό 1 εν γέννη είμαστε σύμφωνοι. Στο project by project ε, είχαμε προτείνει από το άλλο 100.000, 30.000 βλέπουμε εδώ, αλλά φαντάζομαι ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις βλέπουμε ικανοποίηση ότι πολλές φορές ρητά αναφέρονται συμβαστικές τροπολογίες. για την ηλεκτρονική λογοδοσία ε, νομίζω ότι υπάρχει εδώ η κύρια διαφορά μεταξύ της οδηγίας για τη διαφάνεια και της οδηγίας για το accounting, για τα λογιστικά βιβλία. Δηλαδή Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι, ουσιαστικά οι επιχειρήσεις, χωρί εξαιρέσει ή σχεδόν καθόλου, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Και στην έκθεση για το accounting πιστεύω ότι θα πρέπει όχι μόνο σε αιτιολογικές σκέψει, αλλά και στο διατακτικό να μπει η παρατήρηση αυτή για να περάσει στο νομοθετικό κείμενο. Η υποχρέωση για ηλεκτρονική κατάθεση στοιχείων, ανεξαρτήτως όμως του τι τελικά θα κρυφθεί ως προσφορότερο αν θα είναι το XPRL ή κάτι άλλο, γιατί δεν έχω εγώ ιδιαίτερη προτίμηση ενδεχομένω να βρεθεί κάποιο άλλο ευρωπαϊκό πρότυπο πιο χρήσιμο, πιο πρόσφορο. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα να βγει από την αιτιολογική σκέψη και να πάει καλύτερα στο διατακτικό και η προθεσμία του 2018 ίσως θα μπορούσε και να παραταθεί περισσότερο, δεν ξέρω. Συμβαστική 6. Έχω μια ερώτηση για την εισηγητρία. Είχε επαληφθεί η προθεσμία για το πότε θα είναι δημόσιες αυτές οι εκθέσεις πεπραγμένων. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι υπάρχουν ε, επιχειρήσεις οι οποίες, ε, για τις οποίες μαθαίνουμε στοιχεία με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Η σε παραδείγματι, εδώ και 160 χρόνια δραστηριοποιείται στην Κίνα, από το 19ο αιώνα. Ε, δεν θα έπρεπε να είναι κάπως πιο πρόσφατα τα στοιχεία, πιο επίκαιρα και θα έλεγα ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια προθεσμία για το μέχρι πότε πρέπει να διατηθούν ή να μπουν στο διαδίκτυο τα στοιχεία κτλ. Αν περιμένουμε 100 χρόνια για να δοθούν στη δημοσιότητα. Αυτά για τι συμβαστικέ τροπολογίε, της κυρίας Μακάρτη. Καταρχάς, για τον κύριο Λένε τώρα και τι συμβαστικέ του τροπολογίες, πρέπει να πω ότι συμφωνώ εν γέννη, αν και λυπούμε διότι δεν βλέπω αυστηρίο διαχωρισμό μεταξύ του ε, παραδοσιακού, της παραδοσιακών λογιστικών βιβλίων, του accounting του παραδοσιακού και του EFS. Εν πάση περιπτώσει όμως, ε, ίσως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πιο χρήσιμο αυτό. Και αν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, ας είναι, έστω. Σημαντικό επίσης, συμβαστικές τροπολογίες 15 και 16 16 να έχουμε τη νομική βάση για τους μουσουλμικούς ελεγκτές, ώστε και για το μέλλον να υπάρχει αυτή η δυνατότητα επαλήθευσης. Πάλι κοιτώντας και προς το μέλλον και ενδεχομένες τροποποίησεις στη συνέχεια εισαγωγή νέας νομοθεσίας. για τις μικρές επιχειρήσεις ε, και τον δημοσιονομικό έλεγχο. Ε, έκανα διάφορες, είχα διάφορες συνομιλίες και μαθαίνω ότι πράγματα τα οποία ε, σε ορισμένες χώρες για μικρές επιχειρήσεις ελέγχονται μέσω του δημοσιονομικού ελέγχου. Στη Γερμανία, φερειπίνει το ελέγχει ο έφορος απευθείας. Δεν ξέρω αν πρέπει να παρεύουμε σε αυτό το επίπεδο, γιατί αν στη Γερμανία ελέγχει ο έφορος μπορεί στο Βέλγιο από ό,τι μαθαίνω να ελέγχει ένα δικηγόρος τα βιβλία, άρα ίσω δεν χρειάζεται περαιτέρω παρέμβαση στην υπόθεση αυτή. Στο δευτερονικούμενο σημείο που είναι το country by country, Ξέρω ότι έχει κάνει συμβαστικέ τροπολογίε εδώ ο εισηγητή μα και πρέπει να τις συζητήσουμε. Η γραμμή τη ομάδα μου είναι ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα, τη Άλντε. και πολύ διαφορετική από τις συμβαστικές τροπολογίες. Δεν θέλουμε να περιοριστούμε μόνο στην εξορρεκτική βιομηχανία πρώτων υλών ε, και την δασοπονία, αλλά σε όλους τους κλάδους της ε, παραγωγής, ε, της βιομηχανίας. Και βέβαια αυτό πρέπει να το δούμε και σε σχέση με την οδηγία για τη διαφάνεια. Η δε υποχρέωση λογοδοσίας θα πρέπει να αφορά τις επιχειρήσεις άνω των 100.000 ευρώ και όχι των 500.000 ευρώ. Για δε το μέγεθος επιχειρήσης, αν κατάλαβα καλά, μένουμε σε όσα έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι. Πολύ καλά, σε αυτό συμφωνούμε. Συμβαστική τροπολογία, επίσης, ε, η συμβαστική τροπολογία προτείνει μια ημερομηνία εκκίνησης για την υποχρέωση σε περίπτωση που μπορεί να μετατραπεί σε ποινικό αδίκημα μία πράξη σε τρίτη χώρα. Άρθρο 36 και 38 περιγραφή της υποχρέωσης λογοδοσίας effective weight to be applied, χρησιμοποιώ την αγγλική διατύπωση. Και στο 39 βλέπω ένα μικρό πρόβλημα ότι η μητρική εταιρεία που έχει δραστηριότητες ε, στον κλάδο των πρώτων υλών και τον εξορεκτικό και επίσης έχει θηγατρική δραστηριοποιούμενη στον ίδιο χώρο. Και εδώ βλέπω το εξής, ότι ολόκληρος ο όμιλος έχει περιοριστεί μέσα σε ένα ε, τομέα, φερειπίν τον εξορρυκτικό ή των ε, πρώτων υλών, έχει, ε, παρουσιάζει προβλήματα, άρα επηρεάζεται ολόκληρος ο κλάδος, οι και οι θηγατρικές. και προκειμένου να αποφύγει προβλήματα, πολλέ φορέ, γιατί το είδαμε αυτό με αρκετέ ευρωπαϊκέ επιχειρήσει μπροστά στον κίνδυνο των κινέζικων ε, ε, Κινέζων ανταγωνιστών τους ενώ είχαν στο παρελθόν τακτικά προμηθευτεί πρώτες ύλες στην παγκόσμια αγορά αγοράζουν δικές του, δικά τους ορυχεία ε, είτε οπουδήποτε του κόσμου μέχρι και στην Αυστραλία προκειμένου να έχουν μια ελάχιστη διασφάλιση της προμήθειας σε πρώτες ύλες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε. Ένα όμιλο μπορεί να έχει μια διαφορετική κατάσταση για τη Siemens Φερρυπίν, η οποία δεν είναι ε, δε, επιχείρηση εξόρισης πρώτων υλών. Ίσως θα είναι δύσκολο να αντιληφθεί γιατί ρητά αυτή η οδηγία για το accounting μιλάει για ε, πρώτες ύλες και εξόριξη. Ίσως εκεί πρέπει να διαφοροποιήσουμε κάπως το κείμενο. Η κυρία Μακάρτη έχει το λόγο. Συμφωνώ με την κυρία Τάιρα. Πρέπει να ασχοληθούμε λεπτομερώς με αυτούς τους συμβιβασμούς. Είναι σύνθετη η τομή αυτή. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή που έκανε όλες αυτές τις αλλαγές λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες. Τώρα υπάρχουν θετικά στοιχεία τα οποία θα ικανοποιήσουν την ομάδα μου όσον αφορά τον, τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχετε δεχθεί τις ε, τροπολογίες κυρίας Κάστακ του κυρίου Ραγκό. Ε, είναι πολλά τα θετικά στοιχεία, αλλά λόγω πίεσης του χρόνου δεν θα αναφερθώ στα θετικά και ε, δεν θα πω τι, τι μας αρέσει, θα επικεντρωθώ σε αυτά που θεωρούμε ότι, υπάρχουν, ε, ότι έχουν ακόμα προβλήματα. Αυτό αφορά τι διαφορέ μα ε, όσον αφορά τις, ε, τη λογοδοσία της ε, εκθέσεις αναχώρα. Είπατε ότι θέλαμε να ελέγξουμε, να γίνει εναρμονισμό των ετησίων ισολογισμών και ότι αυτό θα, πέσει, θα ξεπεράσει το οικονομικό έτος. Αυτό είναι λογικό. Το θέμα όμως ότι το λογικό είναι υποκειμενικό και αυτό που είναι λογικό για κάποιους δεν είναι λογικό για κάποιους άλλους. Πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε αυτό, να το δουλέψουμε. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και γι' αυτό θέλουμε να συνεργαστούμε για να βελτιωθούν κάποια από αυτά τα ζητήματα. Η δυσκολία που έχουμε με την αναφορά αναχώρα είναι είναι θεμελιώδης και για μένα δεν αποτελεί συμβιβασμό. Δηλαδή, είπατε ότι αν κάποια χώρα συμμετέχει κάποια εταιρεία συμμετέχει σε μια αντίστοιχη ε, απέτηση αναφοράς όπως το ITI θα εξαιρείται αν ήμουν εγώ εταιρεία θα έτρεχα, θα έσπευδα να κάνω ε, να ε, συνταχθώ με ένα τέτοιο σχήμα και, αλλά οι άλλοι θα λέγανε να πάω σε ένα θελούσιο σχήμα αλλά βεβαίως και αυτά λειτουργούν σε κάποιες περιπτώσεις αλλά δεν είναι αντίστοιχα, δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε, που δεν είναι τρόπο να τα θεωρήσουμε αντίστοιχα και έχω δει τέτοιε εκθέσει. και πολύ συχνά, σπανίως μάλλον, ε, ε, ε, δημοσιεύονται και δεν μπορεί κανείς να συγκεντρώσει Λοιπόν, μας ανησυχεί το γεγονός ότι λέμε ότι μπορεί να γίνει κάτι όχι τόσο αυστηρό εθελοντικά. Γιατί λοιπόν τότε χρειάζεται υποχρεωτική νομοθεσία αν μπορεί κανείς να απαλλαγεί ε, εντασσόμενο σε κάποιο εθελοντικό σχήμα. Ίσως να υπάρχουν άλλοι τρόποι να το αντιμετωπίσουμε αυτό, πάντως αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε ως συμβιβασμό, επουδενή. Επίσης, προσπαθήσατε να κάνετε συμβιβασμό στο θέμα της, ε, των εκθέσεων για τις χώρες που ε, ε, ε, ε, υπάρχει αυτή η ιδέα του grandfather clause. Δύσκολο αυτό, γιατί λέτε ότι αν δεν υπάρχει τέτοιος νόμος, η... τι θα γίνει με τη δημοσίευση της οδηγίας στην επίσημη εφημερίδα. Το θέμα που έχω εγώ είναι, ποιες είναι οι χώρες που έχουν κάποιο ποινικό δίκαιο που να ισχύει και να τις αναφέρουμε στο παράρτημα. Αυτή τη στιγμή, καθώς τώρα θα ετοιμάζουμε. Ας μην περιμένουμε ε, για αργότερα που θα εισάγουν τέτοια, θα δούμε τι θα κάνουν. Και αυτό σημαίνει ότι σε κάποια κράτη-μέλη οι, οι τρίτες χώρες που είναι, υπάρχει διαφθορά θα, λένε, θα πούν θα εισάγουμε μια τέτοια νομοθεσία. Και χαίρομαι που έχουμε λίγο χρόνο από αυτού ε, κύριε Πρόεδρε, γιατί το SCC έχουν απαιτήσει στον τομέα αυτό που έχουν εξαιρέσει λόγω της ποινική νομοθεσίας πρέπει να τους δώσουν τα παραδείγματα όπου υπάρχει. Δηλαδή δεν αρκεί να λέει κανεί θέλουμε εξαίρεση. Το ερώτημα είναι γιατί και πρέπει να αποδείξει ότι λειτουργεί σε μια χώρα που σε εμποδίζει να τα εφαρμόσει αυτά. Πρέπει να το κάνουν αυτό, ιδάλλως να πούμε ότι θα έχουμε ένα, ένα παράρτημα, όπου υπάρχει, για να ξέρουμε πού υπάρχει τώρα τέτοια νομοθεσία. Χαίρομαι όπως είπα που υπάρχει χρόνος γιατί θα συναντηθώ με την SCC και για το θέμα της διαφάνειας, αλλά θα φέρουν τους κανόνες 24 Αυγούστου και έχουμε χρόνο να δούμε ποιοι είναι οι δικοί τους κανόνες. Έχω κάνει μια ανταλλαγή απόψεων, άρα θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κατάσταση των καθυστερήσεων. Τους είπα ε, να, δούμε, να δείτε τι θα κάνουμε εμείς και ενδεχομένω να έχουμε εμείς πιο αυστηρούς κανόνες. Ίσως είναι σημαντικό να μην το πιέσουμε αυτό πολύ. Τώρα για τα όρια και τα λοιπά, τα νούμερα, μπορούμε αυτό να το πραγματευτούμε. Υπάρχει περιθώριο εδώ. Θεωρώ όμως ότι από τη σκοπιά τη δική μας θέλουμε να υπάρχει καλός ορισμός του έργου, είναι αδύναμος. Είναι αδύναμο το κείμενο του Συμβουλίου, εσείς κάτι κάπως το προωθήσατε, εμείς θέλουμε ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση και όπως σας είπα ας ασχοληθούμε με το να μελετήσουμε τους συμβιβασμούς, να δούμε τι, πώς μπορούν να βελτιωθούν. Ακούγοντας τις παρεμβάσεις, ξέρω που υπάρχει η πλειοψηφία επ' αυτού στην Επιτροπή μας και ξέρω ότι ποια θα είναι η πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Αν δεν τα βελτιώσουμε αυτά τώρα εδώ, θα μας ε, ε, κατηγορήσουν εξωτερικά ότι, δεν, ότι κάναμε συμβιβασμούς όπου υπήρχε πλειοψηφία για κάποια ισχυρότερη, αυστηρότερη θέση. Λοιπόν, περιμένω τη συνεργασία μας, προσβλέπω σε αυτήν, προοδεύουμε και χαίρομαι γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποια μια συζήτηση όπου είναι αλληλεμπλεκόμενα τα δύο θέματα. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ ε, μιλάει για το accounting, ενώ έχω αναλάβει το θέμα της διαφάνειας, άρα θα μιλήσω πρώτα εγώ για την οδηγία για τη διαφάνεια και μετά θα μοιραστούμε τη συζήτηση με την κυρία Λίχτενμπέργκερ. Εγώ θα περιουστώ σε κάποιες βασικές ε, τοποθετήσεις μόνο. Εν γέννη, Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά ταυτόχρονα και μια πολύ μεγάλη υποχρέωση για περισσότερη διαφάνεια και σαφήνεια για κάθε ένα εμπλεκόμενο στα δικασίε αυτέ. Είτε πρόκειται για τον επενδυτή, είτε πρόκειται για την επιχείρηση που θέλει να είναι σοβαρή, που θέλει να έχει διαφανεί δραστηριότητε για τι κυβερνήσει, για τα κράτη, για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία να θεσπίσουμε κάτι που θα καταπολεμήσει την τόσο αγαπητή αυτή πρακτική της φόρο αποφυγής των ε, μεγαλύτερων συνήθως επιχειρήσεων που μπορούν με διάφορα λογιστικά κόλπα μεταθέτοντας ε, ε, από την μία θηγατρική στην άλλη ή στη μετρική τα λογιστικά στοιχεία να αποφεύγουν την πληρωμή φόρου. Οδηγία λοιπόν για τη διαφάνεια και πεδίο εφαρμογής. Έχουμε διεξοδικά συστήσει το θέμα αυτό. Έχουμε κάνει συστήσει με του κοιόδη έχουμε δει τι τροπολογίε, έχουμε μελετήσει την υπόθεση και μπορούμε να πούμε ότι πολλά από τα σημαντικά θέματα που εμεί τουλάχιστον κρίναμε σημαντικά έχουν καλυφθεί πιστεύω από τι συμβαστικέ τροπολογίε του εισηγητή και τη εισηγητρία. Γι' αυτό και θέλω, θέλω και του δύο να σα ευχαριστήσω. Πρόκειται για μια πολύ καλή δουλειά δώσατε το χρόνο να καθίσετε με τους ε, εμπλεκόμενους με τους σκιώδεις ηγητές, να συζητήσετε, να ακούσετε, να εξηγήσετε, να δείτε τι είναι συμβατό και μη μέσα στο κείμενο. Αυτό όμως που με απασχολεί με ένα περισσότερο είναι να έχουμε δύο ε, εκθέσεις οι οποίες μπορεί εσωτερικά να παρουσιάσουν συνοχή αλλά μεταξύ τους δεν έχουν συνοχή και συμβατότητα και γι' αυτό πρέπει, αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε να έχουμε ένα καλό σύνολο νομοθετημάτων ένα δίκαιο δηλαδή που στο σύνολό του να είναι πρακτικό, να είναι εφαρμόσιμο, να είναι βανάγνωστο και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε σε ορισμένα κεντρική σημασία ζητήματα να δώσουμε κοινού ορισμούς συμμετρικά ούτως υπήν να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια κέρια ζητήματα. Αυτό μπορεί να είναι μια λύση νομίζω. Ιδάλλως, κινδυνεύουμε αντί για σαφήνεια να εισαγάγουμε σύγχυση. Εν γένει. Για τις συμβαστικές τροπολογίες για τη διαφάνεια δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Εγώ δεν έχω προβλήματα. Εν γέννη μα ικανοποιούν και δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Κυρία Λίχτινμπέργκερ, τότε ας περάσω εγώ στο βαρύ πυροβολικό. Ξεκινώ όμω. από τα τελευταία λόγια του, του συναδέλφου ότι δηλαδή πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε να κάνουμε με ένα γενικότερο πλαίσιο και ότι θα χρειαστεί στο συγκεκριμένο, στους συγκεκριμένους τομείς να έχουμε τουλάχιστον συμβατού ορισμού, συμβατή προσέγγιση και μεθοδολογία ώστε να μην ανατραπεί η ασφάλεια και η ισορροπία του δικαίου. Αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερω. επίση θα ήθελα να αναφερθώ και στη γνωμοδότηση τη Επιτροπή των Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων που έχει κάποια σχετικά στοιχεία για το κεφάλαιο υπαριθμών 9. Θέλω να αναφερθώ και να υπογραμμίσω ορισμένε ε, λεπτομέρειες που ίσως χρειάζεται προς συζήτηση. Ορισμός του έργου ή του project. Εάν ε, ακολουθήσουμε τον εσωτερικό ορισμό της επιχείρησης, δηλαδή κινδυνεύουμε να πέσουμε σε παγίδες. Και δεν το θεωρώ σκόπιμο. Πρέπει να έχουμε μια ενιαία αντίληψη, μια σαφή εικόνα του τι σημαίνει project και άρα δεν μπορούμε να εξαρτηθούμε μόνο από τον ορισμό που δίνει η ίδια η επιχείρηση. Και ναι, βεβαίω δεν έχω αντίρρηση να ακολουθούμε θετικέ εμπειρίε και προσεγγίσει που ήδη έχουν ε, εισαχθεί, που χρησιμοποιούνται, αλλά όχι σε αυτό, όχι στον ορισμό. Για το πεδίο εφαρμογή. Ναι, έχουμε διαφορετική αντίληψη για το πράγμα αυτό. Εάν θα έχουμε μόνο την εξόριξη και την δασοπονία ή θα επεκταθούμε και στις λοιπές δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα. Ε, πιστεύω ότι το σωστό θα ήταν να συμπεριληφθεί ολόκληρος ο κλάδος των δραστηριοτήτων μέσα στην έκθεση. Εν τω μεταξύ βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές, ε, πολλές επιχειρήσεις, όμιλοι επιχειρήσεων καλύτερα, με μικτές δραστηριότητες. Ε, αφενός, αφετέρου δεν μπορεί να δοθεί εντύπωση ότι προβάλλουμε κάποιους και ξεχνάμε κάποιους άλλους. Επίσης, συμβαστική τροπολογία για το, που ξεκινάει με το mining and forestry, αλλά στη συνέχεια με την εξόριξη και τη δασοπονία, δηλαδή στη συνέχεια ανοίγει μια θύρα για διαφορετικές λύσεις. Εκεί μπορώ να δεχθώ ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση, δηλαδή να εισαγάγουμε μια ρήτρα που θα δίνει μια διαφορετική προοπτική ε, για το μέλλον. Αυτό θα είναι τουλάχιστον καλύτερο από ότι αυτό που ε, βλέπω τώρα, δηλαδή να περιοριζόμαστε μόνο σε δύο συγκεκριμένου τομεί. Προτεραιότητα για μένα είναι πάλι να ανοίξει το πεδίο εφαρμογή. Στις πληρωμές, το payments. Θα ήθελα πιο πολλές πληροφορίες. Πρόσθετες πληροφορίες σε παραδείγματι που είναι πολύ ενδιαφέρουσες ε, και συναρπαστικές τα πριν το φόρο κέρδη και εν γέννη ο κύκλος εργασιών ε, έχει σημασία να μπουν μέσα στο κείμενο οι οριακές αξίες για 100.000 ευρώ, για 100.000 ε, νομίζω ότι μπορούμε να το δεχθούμε και σαν σημείο σε αυτό να μας οδηγήσει σε μια καλή και λογική λύση για τα reports, για τις εκθέσεις και θα συμφωνήσω εδώ με την κυρία Μακάρτη. Εάν λέμε ότι όποιος θέλει εκούσια μόνο εντάσσεται σε ένα σύστημα reporting, τότε νομίζω ότι έχουμε ουσιαστικά ανοίξει την πόρτα για ε, εικονικές δηλώσεις, ε, για ε, επικάλυψη και στάχτη στα μάτια. Τα έχουμε δει αυτά και στο παρελθόν. Το ε, τις διάφορες εκθέσεις ε, περί κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων που τα γνωρίζω και αρκετά καλά προσωπικώς ε, και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι με καταπλήσει ο τρόπος με τον οποίο μάλλον φιλολογία κάνουν παρά έκθεση πραγματικότητας στον τομέα τη επιστημονική φαντασία κινούνται μερικέ φορέ και νομίζω ότι τη λογοτεχνία πρέπει να την αφήσουμε σε άλλου. Και να έχουν και δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία. Όχι όμω το reporting. Α είμαστε προσεκτικοί. Και α μην ανοίξουμε θύρες που θα μας οδηγήσουν σε εικονικέ ή πλασματικές δηλώσει. Α πούμε ότι δεχόμαστε το σύστημα ΑΜΟΕΣ ή ότι έχουμε τον τάδε κλάδο του εσωτερικού ε, της εσωτερικής λογιστικής, του εσωτερικού reporting, αλλά ας διαλέξουμε κάτι. Ας μην αφήσουμε κάτι το οποίο είναι ε, σε θελοντική βάση να μας παρασύρει σε μη ρεαλιστική καταγραφή στοιχείων. Στη τελευταία ανάλυση όταν έχουμε μια έναν όμιλο κατακαιρματισμένο σε διάφορα κράτη και τμήματα και θηγατρικές δεν μπορεί ο πιθανός επενδυτής να τα παρακολουθήσει όλα. Ε, ας μην παρασυρθούμε λοιπόν στο χώρο της φαντασίας. Πολλά άλλα θα ήθελα να παρατηρήσω, αλλά βλέπω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πάντως είναι ενδιαφέρον ε, Κάτι γίνεται, Α κοιτάξουμε και νομίζω ότι με λίγη προσπάθεια μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό. Ευχαριστώ Επιτροπή. Θέλετε να πείτε τίποτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα σχόλια και από μένα. Ξέρω ότι έχει περάσει η ώρα. Μερικές παρατηρήσεις για την οδηγία για τη διαφάνεια καταρχάς. Μα ικανοποιεί πολύ το συμβιβαστικό κείμενο το οποίο πρότεινε ο εισηγητής. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ θετική η έκθεση. Ε, υπάρχουν βέβαια ένα-δύο πράγματα ακόμα να συζητήσουμε, αλλά μπορεί να γίνει αυτό και ε, σε κατοπινό στάδιο, στους τριμερείς διαλόγους. Όπως σας είπα τώρα για το XPLO, εμείς είμαστε ανοιχτόμυαλοι, θεωρούμε ότι αυτό είναι το μέλλον μας. Ε, θέλουμε να προχωρήσουμε προσεκτικά και με την... Ε, ΕΣΜΑ και δεν νομίζουμε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η ΕΜΣΑ είναι αυτή η οποία θα πρέπει να κάνει τους επιτόπου ελέγχους και τις αξιολογήσεις. Αυτοί είναι άλλωστε οι εμπειρογνώμονες. Αλλά ως προς τη διαφάνεια νομίζω ότι η έκθεση αυτή έχει κάνει τεράστια άλματα. Ε, αφήνω έξω το θέμα της ε, έκθεσης αναχώρα. Ε, όσον αφορά τώρα ε, τις οδηγίες για τα λογιστικά, νομίζω ότι ε, εσείς κύριε Πρόεδρε ως εισηγητές έχετε βελτιώσει αρκετά από τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν. Υπάρχουν βέβαια ακόμα κάποια θέματα προς τη ζήτηση, ιδίως ε, η τροποποίηση του άρθρου 7, ε, εναλλακτική βάση μέτρησης της δίκαιης τιμής και εσείς θέλετε να ε, φύγετε από το μοντέλο που χρησιμοποιούμε μέχρι τούδε. Δεν ξέρω γιατί θέλετε να το κάνετε αυτό αλλά σε μια προηγούμενη τροπολογία η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο μαζί ε, είχαν εισαγάγει αυτή την αλλαγή γιατί ήθελαν περισσότερη ευελιξία ε, για τα κράτη-μέλη και τις επιχειρήσεις. Ε, εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι μέσω αυτής της τροπολογίας χάνεται η ευελιξία που είχαμε προσδώσει το κείμενο στο παρελθόν. Όσον αφορά τις ε, αναχώρα εκθέσεις, να σας το θέσω αλλιώς η πιστοποίηση στις οδηγίες για τα λογιστικά και η οδηγία για τη διαφάνεια, αν δεν υπήρχε ήδη, ε, θα ε, το ολοκληρώνουμε αυτή την εβδομάδα. Η απλούστευση είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις μας. Η έκθεση αναχώρα ουσιαστικά ε, είναι όμοιρος αυτών των δύο προτάσεων διαπιστώνουμε ότι το Κοινοβούλιο αλλά και όλες οι πλευρές επιτυγχάνουν πρόοδο και προσπαθούν ε, να συναντηθούν κάπου και υπάρχουν και κάποιες ε, αρκετά εφάνταστες ιδέες ε, και εμείς θέλουμε να σας διευκολύνουμε εσά και να σας βοηθήσουμε και εσά εδώ στην Επιτροπή ήδη για να βρούμε καλύτερους ορισμούς. Ωστόσο, δύο πράγματα νομίζω ότι πρέπει να έχουμε σαφώς κατά νου. Το πρώτο είναι το πεδίο εφαρμογής. Το πεδίο εφαρμογή ε, των εκθέσεων αναχώρα που ε, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορούσε σαφέστατα την, την βιομηχανία. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το κατάλληλο πεδίο εφαρμογή και θα ε, οδηγήσει σε ισότιμου όρου ανταγωνισμού και ω προ τη ΣΥΠΑ. Ξέρω ότι κάποια κράτη-μέλη θέλουν να προχωρήσουν περαιτέρω και να το εφαρμόσουν για όλε τι επιχειρήσει ή για όλε τι μεγάλε επιχειρήσει τουλάχιστον. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε έναν εντελώς διαφορετικό αντικειμενικό σκοπό και αυτό είναι ε, καταρχάς η φοροαποφυγή. Ε, κανείς δεν είναι κατά ε, της φορολόγησης, αλλά θεωρούμε ότι αυτά τα μέσα δεν είναι τα κατάλληλα μέσα για να καταπολεμήσουμε τη φοροαποφυγή, την ε, φοροαποφυγή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα κάνει μία άλλη πρόταση στη διάρκεια του έτους για να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε τη φοροαποφυγή και τους φορολογικούς παραδείσους θα περιλαμβάνει στο κείμενο, αλλά δεν θεωρούμε ότι το θέμα το των αναχώρα εκθέσεων είναι χρήσιμο σε αυτή την περίπτωση. Το θέμα είναι κατά πόσον επιτυγχάνεται ο στόχο μας. Εμείς κάναμε μια αξιολόγηση αντικτύπου, κάνετε στις συζητήσεις για τις αξιολογήσεις. Ε, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι θα ήταν μάλλον δαπανηρό για τους ε, βιομηχανικούς μας κλάδους, δεν θα ήταν πολύ αποτελεσματικό και θα είναι και ει βάρο τη ανταγωνιστικότητά μα. Αυτά είναι λοιπόν ε, στοιχεία τα οποία αν θέλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη της τη αντικτύπου θα πρέπει να εξετάσουμε. Όσον αφορά τώρα την υλοποίηση των στόχων και τη συζήτηση ε, για τα ε, έργα που αναλαμβάνονται. Νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι η πρόταση που κάνετε ουσιαστικά ε, θέτει ε, την ουσία αυτού που θέλουμε να επιτύχουμε. Δεν θέλουμε οι επιχειρήσεις να επανεξετάσουν το λογιστικό του σύστημα, θέλουμε να υπάρχει δικαιοσύνη και νομίζω ότι αυτό που προτείνετε εσείς είναι πιο δίκαιο και πιο ακριβές. Επομένως θεωρούμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά τον έλεγχο αυτών των εκθέσεων θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην υπάρχουν ε, ε, αλληλοεπικαλύψεις. Θα πρέπει απλώς να γίνεται μία επαλήθευση. Εάν οι εκθέσεις ε, βασίζονται ή προέρχονται από λογαριασμούς που έχουν ήδη ελεγχθεί, ε, δεν ξέρω αν πρέπει να γίνεται και δεύτερος έλεγχος. Ίσως θα μπορούσε να γίνει μια επαλήθευση, αλλά καλό θα ήταν να είμαστε λίγο ρεαλιστές και να προσπαθήσουμε οι δαπάνες για τις επιχειρήσεις να είναι αρκετά χαμηλές. Μια διαδικασία όμως ελέγχου, πιστοποίησης τουλάχιστον θα έπρεπε να υπάρχει. Ε, τι άλλο, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε. την αξιολόγηση για το κατά πόσον υπάρχει νομοθεσία σε ποινικό επίπεδο. Θα ήθελα να ε, ακούσουμε ένα κατάλογο, να δούμε και τι γίνεται. Ε, ο κλάδος ενδιαφέρεται για το θέμα και έχουμε πάντα το παράδειγμα της Κίνας. Ε, αυτή η ιδέα μιας ε, ρήτρα grandfathering είναι καλή. Ε, θα προσπαθήσουμε όμως να την έχουμε όσο δυνατόν πιο περιορισμένη, διότι δεν θέλει κανείς να ξεπηδήσουν ε, νέες νομοθεσίες οι οποίες ουσιαστικά θα κάνουν ε, ανύπαρκτη την πρότασή μας. Δεν είναι ο στόχος μας αυτός. Θέλουμε να επιτύχουμε, αλλά θέλουμε να γίνει με τον κατάλληλο τρόπο και στον κατάλληλο χρόνο. Να ε, προσπαθήσουμε λοιπόν στις επόμενες εβδομάδες να λύσουμε και τα τελευταία προβλήματα. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Πρόεδρος, μια και δεν έχουμε άλλο χρόνο, δεν θα πούμε τίποτα παραπάνω. Θα κοιτάξουμε το θέμα ταξίς και των εισηγητών. Σεπτέμβριο θα είμαστε έτοιμοι και θα επιδιώξουμε στις αρχές της, εβδομάδα εβδομάδας του Στρασβούργου να προβλέψουμε μια συνάντηση, Δευτέρα ή Τρίτη, όχι προ το τέλο, αλλά στην αρχή μάλλον της, εβδομάδα εβδομάδας του Στρασβούργου. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει οι συνεργάτες μας τεχνικά να έχουν προετοιμάσει τα θέματα ε, την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από το Στρασβούργο δηλαδή. Αφήνουμε το σημείο αυτό και πάμε στο επόμενο θέμα που έχουμε κρεμές και είναι το 36 πρόγραμμα δικαιώματα και ηθαγένεια. Μόνο προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών πρέπει να ορίσουμε. 18 Ιουλίου, αν δεν έχετε αντίρρηση, 37 αναβάλλεται, 38 στα διάφορα, όχι τίποτα, προσεχή συνεδρίωση, 17 και 18 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.